Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε. Ξεκινάει η συνεδρίαση. πριν να δώσω κάποιες διευκρινήσεις, θέλω να ρωτήσω αν έχετε αντιρρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Καταρχάς, δύο προσθήκες. Σας έχουν διανεμηθεί ο κύριος Γκάιερ, υποβάλλει Βράχει πρόθεσμα έκθεση για την ε, κινητοποίηση του contingency margin του περιθωρίου για απρόβλεπτο κομμάτι του πακέτου του, της συνδιαλλαγής για τον προπολογισμό 2018 και ένα κατεπήγον αίτημα με τον αριθμό 33 που στόχο έχει τον περιορισμό του προενταξιακού μέσου για την Τουρκία ε, ε, υπέρ της ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της Συριακής κρίσης. Ίσως εάν ε, μας είχε καταστεί γνωστό την ε, στιγμή της συνδιαλλαγής ε, αυτό το αίτημα μεταφοράς, θα είχε διευκολύνει πολλούς που είχαν κάποιες επιφυλάξεις και ανησυχίες. Εάν δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, το άρθρο 18 πάντως, το σημείο 18, ενημέρωση για τριμερείς διαλόγους, σας ενημερώνω ότι θα έρθει στη συζήτηση στο 5 σήμερα το πρωί. Και το θέμα Κονουσβάν θα πάει αμέσως μετά τις ψηφοφορίες στις 5.30. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις. Ανακοινώσεις. Το σχέδιο αποφάσεων των συντονιστών της 9ης Οκτωβρίου σας έχει κοινοποιηθεί βρίσκεται στο φακελό σας και αν δεν έχετε σχόλιο θεωρείτε πως εγκρίνονται αυτές οι αποφάσεις και δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Η σημερινή συνεδρία ξεκινάει στις 14.30 και καινοτομούμε. Μπορούμε από εδώ και μπρος να αρχίζουμε στις 2.30 και όχι στις 3 όπως συνέβαινε μέχρι τώρα και τελειώνει στις 18 και 30 ακριβώς. Και θα ευχαριστώ τον Hans Γκέιερ, ο οποίος ε, θα προεδρεύσει. Εγώ έχω μια δέσμευση. Γιατί εδώ στι Βρυξέλλες λαμβάνει η χώρα η Skills Week, η εβδομάδα των δεξιοτήτων και μου έχει ζητηθεί να λάβω το λόγο για να αναφερθώ στο πιλωτικό μας πρόγραμμα για την ε, ε, κινητικότητα των ε, ασκουμένων, μαθητευμένων στην Ευρώπη. Τα πρακτικά της 30ης-31ης Αυγούστου και 26ης-27ης Σεπτεμβρίου έχουν κοινοποιηθεί εγκαίρους. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις ή προτάσεις για τροποποίηση, θεωρούμε πως εγκρίθηκαν. αποτελέσματα της συνδιαλλαγής. Συμβούλιο και Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Και υπενθυμίζω ότι επετεύχθη συμφωνία τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, στο πλαίσιο της Επιτροπής της Συνδιαλλαγής, μια συμφωνία η οποία επισφραγίστηκε κάπου στις 4 το πρωί σε προηγούμενη συνεδρία του προπολογισμού πριν από δύο εβδομάδε, οι προοπτικέ ήταν μάλλον ζωφερές. Η Επιτροπή δηλαδή θεωρούσε ότι το δικό της σχέδιο προπολογισμού ήταν το μόνο δυνατό σημείο ισορροπίας μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και ότι ε, αναδιπλώσεις μεταφορές, προσαρμογές που είχαν συμφωνηθεί πέρσι ήταν ένα είδος ιερού και θεόπνευση του βιβλίου, μια βίβλωση η οποία δεν θα μπορούσε να ανατραπεί, δεν θα μπορούσαμε να την ε, ξεχάσουμε, να την ξεπεράσουμε, να την υπερβούμε. Ε, καμία δηλαδή διόρθωση ρύθμιση σε σχέση με το πολιετές πρόγραμμα αυτό ήταν όλα παγιωμένα και εδρωμένα Το Συμβούλιο προχωρούσε σε μια περιοριστική, μια συσταλτική ερμηνεία της ε, μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης και το ενδιέφερε μόνο η διατήρηση περιθωρίων για να αντιμετωπίσει τα λεγόμενα απρόοπτα παράταση λίγο πολύ του λεγόμενου μέσου για τους πρόσφυγες στη Συρία ήταν τα λεγόμενα απρόβλεπτα ε, με μία πρόταση που αρχικά είχε ακουστεί για ένα δισεκατομμύριο, το μεταξύ έχουμε συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη σε επίπεδο τριών δισεκατομμυρίων ε, και μετά θα έρθει άλλο ένα ε, ποσό για το 2018 ε, τα κράτη-μέλη, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το ένα δισεκατομμύριο που έπρεπε να προσφέρουν τα υπόλοιπα δύο αυτή τη στιγμή ε, ψέγονται, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συμμετάσχουν και έτσι θα κληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των δύο δισεκατομμυρίων που λείπουν των τριών συνολικά. Άρα, η προσέγγιση του Συμβουλίου είχε σαν ε, συνέπεια τη διατήρηση ενός περιθωρίου περί τα 3 δις και άρα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν ήταν καν πραγματικός προϋπολογισμός. Διότι δεν ενεγράφοντο εξ αρχής προβλεπόμενες διαπάνες. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή και με τη νύχτα προς το Σάββατο μπορέσαμε να ε, διασκεδάσουμε αυτές τις ανησυχίες και τα εμπόδια μετά την αναγνώριση από πλευρά του Επιτρόπου την ότι ούτε το Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο σεβόνταν κατά γράμμα την κοινή δήλωση για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και ότι ως εκ τούτου ήταν σε θέση ε, η Επιτροπή να εγκρίνει κονδύλια που ε, θεωρούσε σκόπιμα στην ετήσια διαδικασία και επίσης ε, συμφωνήσαμε ότι στη διαδικασία ενίσχυσης του τίτλου 1α έπρεπε να δώσουμε τις πραγματικές ε, προτεραιότητες στο ορίζον 2020 στο έρασμο στο κόσμο που δεν μπορούν να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με αυτό των προθέσεων ή δηλώσεων του Συμβουλίου στο πλαίσιο των ίδιων προγραμμάτων και έτσι εξασφαλίσαμε επιπλέον κονδύλια 105 εκατομμύρια με φρέσκο χρήμα για τον τίτλο 1α κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για την ανάληψη των υποχρεώσεων και επίσης στο 1β είχαμε σημαντική ενίσχυση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. 50% των πιστώσεων που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς πλέον αυτό να θεωρείται προκαταβολή του ποσού που είχε loading, δηλαδή του ποσού που είχε συμφωνηθεί στην ε, διάμεση ε, πορεία. Και είπαμε επίσης ότι το προενταξιακό μέσο για την Τουρκία περικόπτεται με αντισταθμίσμα κατά 85 εκατομμύρια ευρώ ε, ενίσχυση σε άλλα προγράμματα. Το Κοινοβούλιο επίσης ικανοποιείται προς τις τροπολογίες του σε άλλους τίτλους σε σχέση και με τις υπηρεσίες και με ένα πιλωτικό πρόγραμμα δράσης και προετοιμασίας με 100 εκατομμύρια ευρώ και κάτι. Το Κοινοβούλιο επίσης αποκαθιστά το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών που είχε επιβάλει το Συμβούλιο και επίσης οι τροπολογίες που κερδίσαμε εμείς έχουν χαρακτηριστικό σήμα ε, τις επιλογές του Κοινοβουλίου, δηλαδή δεν, χαρακτηρίζονται δεν εισάγονται με διορθωτική επιστολή της Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός, ε, ο απολογισμός μάλλον αυτή ε, στη συνδιαλλαγή για τον είναι γενικά θετικός αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε επιτύχει πολύ σημαντικές επιτυχίες. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή είχαν ε, αντισταθεί με επιχειρήματα επί της αρχής ιδιαίτερα ε, έντονα και για το Brexit και για την ε, μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και για το μέσον για την Τουρκία δεδομένων δε και των υποεκτελέσεων στις πληρωμές το Συμβούλιο ήθελε ιδιαίτερα να πλήξει τις αναλήψεις υποχρεώσεων με δεδομένα όλα αυτά, μπορεί το αποτέλεσμα δεδομένη τη δική μα στράτευση και προσήλωση να μην ήταν αναπάντεχο, αλλά πάντω είμαστε πολύ ικανοποιημένοι σε σχέση με τι προσδοκίε μα, οι οποίε ήταν βέβαια αρκετά μετριοπαθείς δεδομένου ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Δεν θέλαμε να αυξήσουμε δαπάνες διότι η αύξηση δημοσίων δαπανών δεν αποτελεί προσδοκία της ευρωπαϊκής κοινή γνώμη Και έτσι πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι αυτά που προτείνουμε θα αντιστοιχούν και στην προσδοκία του δημοσίου αγαθού που περιμένει η Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη και ότι έτσι θα προετοιμάσουμε το μέλλον της Ευρώπης προσφέροντας ασφάλεια στους Ευρωπαίους. Πολλοί συνάδελφοι διαδραμάτισαν ε, ρόλο σημαντικό στην Επιτροπή της Συνδιαλλαγής, ε, αναπτύσσοντας και ενεργοποιώντας επαφές που έχουν σε επίπεδο κυβερνήσεων κρατών μελών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο για να προετοιμάσουν το έδαφος. Θέλω να τους ευχαριστήσω εδώ ιδιαιτέρως γιατί πρέπει να πω ότι στενόμαστε μια κάποια δυσφορία όταν απέναντί μας έχουμε υπουργούς, λίγοι βέβαια ήταν, κάποιους ε, πρεσβευτές και κάποιους εκπροσώπους μονίμων αντιπροσωπιών που ωστόσο είναι ε, επιτετραμένοι των Υπουργείων Οικονομικών ανώτεροι αξιωματούχοι που όμως έρχονται χωρίς κανένα περιθώριο διαπραγμάτευσης και έτσι αυτό μας φέρνει σε δύσκολη θέση και μας προξενεί μεγάλη δυσφορία μας στους βουλευτές. Ο Επίτροπος Έτεγκερ και το επιτελείο του επίσης αξίζουν συγχαρητηρίων και τι ε, κατά καιρού θεώρησα ότι ήταν κάπως ε, άτοπα κάποια σχόλια σε σχέση με δισταγμούς και επιφυλάξεις που αναγνώριζε σε κάποια κράτη-μέλη καθαρούς ε, Χρηματοδότε του προπολογισμού και ίσω θα έπρεπε να το έχω μιλήσει πιο καθαρά. Επίσης ευχαριστώ τον Υπουργό Κιβεν και την ομάδα της Προεδρίας, τη Γραμματεία του Συμβουλίου που έκαναν πολύ καλή δουλειά τόσο τεχνικού επίπεδου όσο και πολιτικής διαπραγμάτευσης προκειμένου να εξασφαλίσουν διαμεσολάβηση έτσι ώστε να εξασφαλίσουν συμφωνία από θέσεις οι οποίες ήταν διαμετρικά αντίθετες. Επίσης, ο κύριος Σίκφριτ Μουρεσάν, γενικός εισηγητής, έκανε καταπληκτική δουλειά, τη χαιρετίζω εδώ, επίπεδο αριστείας χαρακτηρίζει το έργο του και οφείλω να τον συγχαρώ και να, ε, να σημειώσω πόσο με εντυπωσίασε η αποτελεσματικότητα και η προσήλωσή του στη δουλειά αυτή. Τον συγχαίρω λοιπόν και τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίση και συγχαίρω τον Ρίτσαρντ Άσχουετ, εισηγητή των λοιπόν τμήματων. Δεν ήταν εύκολο το έργο του. Ιδιαίτερα όταν ε, έχει κάνει στα χέρια του ένα τρίτο ε, έγγραφο με περιορισμούς για τις πιστώσεις σχετικές με τα κτίρια. Σε ευχαριστώ, Ρίτσαρτ. Τον εισηγητή τον αρμόδιο για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες Ρίχαρτ Γκέιερ και για τον προπολογισμό βέβαια 2017 έδειξε αιμονή, επιμονή και μεγάλη δυνατότητα ισορροπίας και ισορροπισμού. Ε, επίσης περιμένουμε του, τώρα ο εισηγητής να μας κάνει την παρουσίαση του για τις ε, εντυπώσεις του από αυτή τη διαδικασία του συνδιαλλαγής και δίνω το λόγο ανευπεραιτέρω στον κύριο Μουρεσάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς από εσά ε, μετά από τόσες ώρες, ε, έχοντας περάσει τόσες ώρες μέχρι το Σάββατο το πρωί στην συνδιαλλαγή. Πρώτον, επειδή η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον πρόεδρο Αρτουή που έπαιξε τόσο σημαντικό και ενεργό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της συνδιαλλαγής. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο διότι μας ε, ε, έδωσε τη δυνατότητα να φτάσουμε σε αυτή την πολύ καλή συμφωνία επί του προϋπολογισμού με το Συμβούλιο, θεωρώ. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής μας ε, και αυτοί ε, δούλεψαν άοκνα τις τελευταίες εβδομάδες, ήταν πάντοτε στο πλευρό μας ε, κάθε φορά που χρειαζόμασταν πάντα με αφοσίωση και επαγγελματισμό όπως και με δημιουργικότητα μας υποστήριξαν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για το έργο τους τους δύο εισηγητές με τους οποίους εργάστηκα πιο στενά, τον Ρίτσαρτ που ήταν υπεύθυνο ε, για, για τα άλλα κεφάλαια και τον κύριο Γκάιρ που ήταν υπεύθυνο για τα Στου ε, αποκεντρωμένους φορείς ε, ήταν και γενικός εισηγητής για το 2017 οπότε η συνεισφορά του ήταν πολύ σημαντική αποτέλεσε σημαντικό πυλώνα των διαπραγματεύσεων και της συμφωνία. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Έτιγκερ ο οποίο δεν είναι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή όμως εκτιμώ ιδιαίτερα. Επίσης το ε, προσωπικό της DG Budget ήταν, ήταν στο πλευρό μας, βρήκανε λύσεις, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη συνδιαλλαγή. Τώρα σύντομα θα σας περιγράψω περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η συμφωνία, γιατί θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι καλός. Όπως είπα, στο τέλος της συνδιαλλαγής στις 3.30 το πρωί ε, ζήτησα από τους συναδέλφους ε, του Κοινοβουλίου να αποδεχθούν και να εγκρίνουν αυτόν τον προβλέψιμο στον ε, κεφάλαιο 1α. Έχουμε 105 εκατομμύρια φρέσκου χρήματος για τις προτεραιότητές μας αυτούς τους τομείς. 17 εκατομμύρια για τον ορίζοντα 2020, 20 εκατομμύρια για το Εράσμους και 15 για το Κόσμε αυτή ήταν μία από τις top προτεραιότητες του Κοινοβουλίου γιατί μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φοιτητέ, την έρευνα και την ανάπτυξη. Είναι οι τομείς ε, όπου χρειάζονται χρήματα, όπου δαπανώνται σωστά και ε, κάνουν την Ευρώπη πιο προσανατολισμένη προς το μέλλον. Όπως σας είπα είναι φρέσκο χρήμα, δεν υπάρχει ανακατανομή, δεν υπάρχουν ε, υποσημειώσεις και αστερίσκοι ε, που να λένε ας πούμε ότι η αύξηση φέτος πρέπει να αντισταθμιστεί του χρόνου. Είναι ξεκάθαρη ε, νίκη 105 εκατομμυρίων φρέσκων πιστώσεων. Τώρα, στο 1β η ανεργία των νέων. Αυτό ήταν μια προτεραιότητα της πλειοψηφίας των μελών ε, του σώματος και πολλών πολιτικών ομάδων. Ο Επίτροπος βάσει της ε, περσινής συμφωνίας είχε προβλέψει 233 εκατομμύρια για την ανεργία των ε, νέων. Είπαμε ότι δεν αρκούν και καταφέραμε να έχουμε 116 εκατομμύρια ευρώ σε φρέσκες πιστώσεις. Είναι αύξηση κατά 50% ε, είναι φρέσκα χρήματα, δεν είναι μπροστοβαρής η επιβάρυνση όπως ήθελε το Συμβούλιο και είναι ξεκάθαρη νίκη για το Κοινοβούλιο. Ε, επίσης έχουμε μία κοινή δήλωση Συμβουλίου, ε, Κοινοβουλίου και Επιτροπής που λέει ότι αν χρειαστούν περισσότερα χρήματα για την ανεργία των νέων θα διατεθούν. Επίσης έχουμε και τα ποσοστά απορρόφησης φέτος. Αν απορροφηθούν όλα φέτος θα έχουμε και του χρόνου κάποια χρήματα ε, σε περίπτωση που δεν δαπανηθούν φέτος. Κατάλαβα στις διαπραγματεύσεις ότι η δέσμευση του Επιτρόπου είναι ξεκάθαρη. Θέλει να ενημερώνει το σώμα ως προς τις ανάγκες επιτόπου και σε περιοδική βάση του χρόνου, έτσι ώστε του χρόνου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ε, κατά πόσο χρειάζονται περισσότερα και αν χρειαστούν να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε με τα σωστά στοιχεία. Δεν υπάρχουν λοιπόν αστερίσκοι ούτε υποσημειώσει με αυτό το φρέσκο χρήμα. Στο κεφάλαιο 2 έχουμε 34 εκατομμύρια ευρώ για του νέου γεωργού. Όπως ξέρετε θέλουμε να κάνουμε περισσότερα για του νέου γεωργού. Η Κομισιόν ήδη αυτό το είχε περιλάβει στην τροποποιητική επιστολή. Καταφέραμε αυτό μέσω τη συνδιαλλαγή να το διασφαλίσουμε χρήμα λοιπόν 34 εκατομμυρίων για τους νέους ε, ε, αγρότες στην ε, κεφάλαιο 3 δεν υπήρχαν περιθώρια όπως ξέρετε οποιαδήποτε αύξηση εκεί πρόκειτο να έρθει από το μέσο ευελιξίας. Καταφέραμε λοιπόν να καλύψουμε τη βασική μας προτεραιότητα της αποκεντρωμένους οργανισμούς του Κοινοβουλίου να πάρουν τα εξής ποσά. πολ 3,7 εκατομμύρια ευρώ και 10 θέσεις. Εάζω 5 εκατομμύρια ευρώ και 1,8 εκατομμύρια ευρώ και 5 θέσεις για τη Eurojust. Νομίζω ότι αυτό είναι καλή ισορροπία και αντικατοπτρίζει και τις πολιτικές προτεραιότητες των ομάδων, των διαφόρων ομάδων στο Κοινοβούλιο. Στο κεφάλαιο 4 καταφέραμε να έχουμε αυξήσει 85 εκατομμύρια ευρώ σε αυτές τις γραμμές που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να ενισχυθούν και αυτές είναι καταρχάς το NSF. 34 ε, εκατομμύρια για το NEAST, e 20 ε, για την ε, εργαλείο ανάπτυξης της συνεργασίας και 2 εκατομμύρια για την στρατηγική συνεργασία για την αντιμετώπιση των στοιχείων από την ε, Ρωσία 2 εκατομμύρια για την τουρκοκυπριακή ε, κοινότητα και 1,5 ε, εκατομμύριο για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. Αυτό και πάλι είναι το ίδιο ποσοστό με αυτό που ζητήσαμε στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. αποφασίσαμε να κόψουμε έτσι φιλόδακτα τα προεντεξιακό μέσο για την Τουρκία. Η θέση μας ήταν να κόψουμε 50 εκατομμύρια και να έχουμε 30 εκατομμύρια σε απόθεμα. Αυτή η φιλοσοφία διατηρήθηκε, οπότε έχουμε και την περικοπή και το απόθεμα, αλλά μαζί με το Συμβούλιο αποφασίσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι, γιατί βλέπουμε τις εξελίξεις στην Τουρκία. Η Τουρκία απομακρύνεται από τα ευρωπαϊκά στάνταρτ σε επίπεδο δημοκρατίας, κράτους δικαίου, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ελευθερίας ε, του τύπου και της έκφρασης. Αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε απαρατήρητο. Έτσι η περικοπή είναι 105 εκατομμύρια ευρώ και το αποθεματικό είναι 17 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που είναι καλό επίσης είναι ότι ε, το απόθεμα αυτό ήταν και η φιλοσοφία του Κοινοβουλίου όπως και η περικοπή γιατί έτσι η κυβέρνηση στην Άνκαρα βλέπει ότι αν ε, βελτιωθούν τα πράγματα θα έχουν χρήματα αλλιώς όχι. Τις πιλωτικές δράσεις ε, δεν το συζητήσαμε ε, στη συνδιαλλαγή γιατί το πακέτο του Κοινοβουλίου εγκρίθηκε όπως και τα προηγούμενα χρόνια χωρίς συζήτηση όμως η διαφορά φέτος σε σχέση με πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι κάναμε πλήρη χρήση των πιστώσεων που ήταν διαθέσιμα ε, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό για αυτό το θέμα. Φυσικά η προπαρασκευαστική δράση για την άμυνα ήταν από το Συμβούλιο και το Κομισιόν δεν ήταν προτεραιότητα του Κοινοβουλίου και έτσι ε, ε, ένα μεγάλο ποσό πηγαίνει προς τα εκεί. Από την άλλη όμως είναι η πρώτη φορά που κάνουμε πλήρη χρήση αυτών των πιστώσεων όπως είπα. Ε, συνολικά να πω το εξής. Όπως ξέρετε, πέρυσι όταν εγκρίθηκε ο προπολογισμό και μέσα στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης είχαμε περικοπές στο κεφάλαιο 1 και το Συμβούλιο είχε θεωρήσει ότι φέτος έπρεπε αυτές να αντισταθμιστούν. Συγγνώμη, οι αυξήσεις διορθώνει ο εισηγητής. Ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ. Η θέση με την οποία ξεκίνησα στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο ήταν ότι αυτοί θεωρούσαν πως έπρεπε να πάρουν κάποιες περικοπές και κάποιες κάποια κράτη-μέλη, όπως και η Προεδρία, μας είπαν ότι πρέπει να κόψουμε 200 εκατομμύρια από, την, ε, από το κεφάλαιο 1. Ε, καταφέραμε να αντισταθούμε σε αυτές τις περικοπές ε, και στο τέλος καταφέραμε να έχουμε και 105 εκατομμύρια σε φρέσκο χρήμα. Καταφέραμε να αντισταθούμε σε όλες τις περικοπές, όπως είπε και ο Πρόεδρος, σε μεγάλο βαθμό καταφέραμε να δώσουμε τη σωστή ερμηνεία στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε η αναθεώρηση, αλλά ήταν ξεκάθαρο και και γραμμένο στο χαρτί ότι δεν πρέπει να προκαταβάλλεται ο ρόλος μας ως δημοσιονομική αρχή. Τις προερασμένες εβδομάδες ήμασταν σε μια θέση με τα χέρια δεμένα και τελικά αν... Ε, θα έπρεπε ε, η τελευταία μας λέξη να ακουστεί για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα για τα, ε, για τα υπόλοιπα κεφάλαια που είχαμε φρέσκο χρήμα είδαμε ότι η δημοσιονομική αρχή δεν έχει περιοριστεί, δεν έχει τελειώσει μέχρι τα τέλη του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό είναι καλά νέα για μένα, για εσάς και για τους συζητητέ τα επόμενα δύο χρόνια. Για να καταλήξω λοιπόν, Θεωρώ πως έχουμε πολύ καλό προϋπολογισμό, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητές μας και νομίζω ότι έχουμε έναν καθαρό προϋπολογισμό χωρίς κρυμμένες βόμβες που θα σκάσουν τα επόμενα δύο χρόνια ε, μέσα στα πλαίσια του πολιετούς. Ε, δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ε, ή παρενθέσεις που θα προκαταβάλουν τα επόμενα έτη τον προϋπολογισμό και θα περιορίσουν την ισχύ της θέσης μας. Γι' αυτό Χαιρόμαστε για τη συζήτηση σήμερα το πρωί και ζητώ κυρίως από τους ε, συναδέλφους από όλες τις πολιτικές ομάδες να υπερψηφίσουν αυτόν τον προϋπολογισμό και αυτά τα συμπεράσματα της συνδιαλλαγής την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια όπου είναι στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω το λόγο στον ε, κύριο Ντεσμέρση, στον κύριο Γεγέρ, στον Γκάιλινγκ στον κύριο Άσφορτ, να συγχωρείτε, ε, στην Γενική Διευθύντρια της Επιτροπής και μετά στους συντονιστές και σε όσους ε, θέλουν να εκφραστούν, να αντιδράσουν σε αυτή την συμφωνία της συνδιαλλαγής. Ο, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να απηχήσω τα σχόλια που κάνατε εσείς και ο κύριος Μουρεσάν μας στιγμή ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικό το αποτέλεσμα και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερο τον Γιάν Σκάιερ και τον Ζήκριτ Μουρεζάν που πιστεύω ότι έκαναν ε, εξαιρετική δουλειά. Θα γνωρίζετε ότι από αυτές τις περιστάσεις και, ε, περιστάσεις και επειδή επιτύχαμε κάποια πράγματα, παρότι είχαμε περιορισμένο ε, περιθώριο λιγμού για το τίτλο 5, πετύχαμε κάποια πράγματα αλλά όχι όλα. Από την άλλη πλευρά, θα, με χαρά μπορώ να σας αναφέρω ότι η αύξηση του 2,5% είναι λογική και αποδεκτή. 800.000 ευρώ για τη δημιουργία ενός, ε, μιας γραμμής για τις στρατηγικές επικοινωνίες δημιουργήθηκε ε, η γραμμή. Ήταν ένα από τα κύρια θέματα που υποστήριξε το Κοινοβούλιο και όλες οι επιτροπές το στήριξαν και από την πρώτη μέρα κερδίσαμε το επιχείρημα. Γι' αυτό και νομίζω αυτό πρέπει να μας ικανοποιήσει. Για τους υπόλοιπους θεσμούς ε, ε, νομίζω πως είχαμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα με δύο απογοητεύσεις. Το πρώτο αφορά το ελεγκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει λογική και αιτιολογημένη ε, αιτιολογημένο αίτημα για αύξηση στον προπολογισμό όμως ε, έμενα με την εντύπωση και κατάλαβα ότι μπορεί και να αναθεωρηθεί και να υπάρξει μια δυνατότητα να συζητήσουμε περαιτέρω τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου, λέει τώρα ο ναι. πω αυτά, εκεί θα χρειαστεί να γίνει κάποιος συμβιβασμός. Και στην τελευταία μου παρατήρηση να πω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, της Διαπραγμάτευσης πρέπει να εξορροπήσει τις απόψεις σε ένα σωρό απόψεις. Πρέπει να εξορροπήσει τις απόψεις ε, των, του Συμβουλίου, των Επιτροπών της Επιτροπής και υπό χρονικό περιορισμό. Δεν είναι καθόλου εύκολη η υπόθεση του Προέδρου της Επιτροπής Προπολογισμού. <coughs> το να λάβεις τέτοιες αποφάσεις 4 το πρωί, ε, νομίζω ότι πιέζει όλους τους διπλωματευτές. Θα πρέπει να σκεφτούμε αυτό το προπολογισμό 60 δις αν χρειάζεται να κάνουμε έξτρα προσπάθεια για ακόμα 5 εκατομμύρια για ένα σχετικά μικρό θέμα. Αυτό ε, ο πρόεδρος θα πρέπει να το σκεφτεί και να το κρίνει ε, και θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο και να το μπροστά σε ολόκληρη την Επιτροπή για το πώς ε, έκανε τις διαπραγματεύσεις εξ ονόματός μας. Θέλω λοιπόν οι ιδιαίτερως να ευχαριστήσω τον πρόεδρο. Ευχαριστώ, Ρίτσαρντ. Το λόγο τώρα έχει ο Γιάννης Γκιάγερ για τους οργανισμούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για τα θερμά συγχαρητήρια, τα ανταποδίδω. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή συνεργασία πάνω από όλα πέραν των κομματικών φραγμών από πλευράς της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Μια πολύ θετική εμπειρία γιατί ξεπεράσαμε τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές ε, και είχαμε πολύ καλή συνεργασία με σταθερές και συνεπείς θέσεις σε όλη τη διαδικασία εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Δεν είναι εύκολο αυτό και νομίζω ότι μας ενθαρρύνει και μας, δίνει, μας δείχνει πώς πρέπει να δουλεύουμε από εδώ και μπρος. Ο Ζίκφριτ βέβαια ανέφερε ήδη τα κύρια θέματα που αφορούν τους αποκεντρωμένους φορείς ή υπηρεσίες. Προτεραιότητα του Κοινοβουλίου, όπως το αναμενόμενο, ήταν, δεδομένου ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση του προσφυγικού. Ε, ιδιαίτερη λοιπόν ήταν η έμφαση για μας στη κατηγορία 3 στις σχετικές υπηρεσίες. Εκεί δώσαμε την έμφαση, εκεί κάναμε την ε, πιο σκληρή δουλειά και μπορέσαμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις να στρέψουμε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και σε οι υπηρεσίες της κατηγορίας 1α, η GSA παραδείγματι που είναι υπεύθυνη για την ε, ε, ε, εκτέλεση του προγράμματος Γαλιλαίος με πολύ μεγάλη σημασία για την καινοτομία και την τεχνολογία στο δορυφορικό αυτό πρόγραμμα που προχωράει και θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί. Οι αποκεντρωμένοι φορείς και υπηρεσίες είναι βεβαίως μικρό κομμάτι του προπολογισμού αλλά πάντα πολύ σημαντικό διότι Εάν ε, έχει κάποια ιδέα για το τι είναι αυτές οι υπηρεσίες, η κοινή γνώμη συνήθως έχει την ιδέα ότι είναι υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός τους. Από την άλλη, όταν πρόκειται να διατεθεί κάποια από αυτές, ε, τα κράτη-μέλη αμέσως διαγωνίζονται για να δούνε ποιο θα καταφέρει να την ε, εξασφαλίσει. Επομένως, σε σχέση με τις υπηρεσίες βλέπουμε να υπάρχει μια όχι πολύ καθαρή στάση από πλευράς των κρατών μελών. Και επίσης σε σχέση με τον προπολογισμό του 2018 έχουν ε, ε, επιτελέσει, έχουν εκτελέσει την υποχρέωσή τους οι υπηρεσίες για περιορισμό του προσωπικού ε, κατά 5% όπως προκύπτει από τη Διοργανική Συμφωνία. Αυτό δεν το δεχόταν το, το Συμβούλιο. Στην προσεχή στις δημοσιονομικές ε, προοπτικές φαίνεται το Συμβούλιο να απειλεί με επιπλέον περικοπές ε, προσωπικού, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε προβλήματα λειτουργικότητας πλέον τους ε, αποκεντρωμένους οργανισμούς αλλά και τα θεσμικά όργανα τα ίδια. Και γι' αυτό και ως ηγετής του 2017 επιτρέψτε μου να πω ότι ο τροποποιητικός του προϋπολογισμός του 2000, Έξι, συμπληρωματικός ε, τροποποιητικός προϋπολογισμός του 2006 ήταν μέσα στο πακέτο στο οποίο εξετάσαμε. Δεν είχαμε χρόνο ιδιαίτερα να συζητήσουμε διεξοδικά τις αποφάσεις. Απλώς επισημάναμε στο Συμβούλιο πώς προχωρούν οι εξελίξεις, πώς προχωρούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, ποιες είναι οι δικές μας οι θέσεις. και καθώς μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε απαντήσεις οι οποίες ήταν αρκετά ικανοποιητικές σήμερα μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε στο διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 6. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του πακέτου μπορούμε να κινητοποιήσουμε τώρα ένα περιθώριο για το οποίο ε, θα συμφωνήσουμε σήμερα στις ε, πρακτικές διευθετήσεις. Για μένα λοιπόν το, το δικό μου μέρος της δουλειάς ως εισηγητή του 2017 έχει λίγο πολύ ολοκληρωθεί, ολοκληρωθεί μια-δυο μικρομεταφορές ε, κονδυλίων. Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Παραδίδω τη σκητάλη στον Ζεκφίτ Μουρεσάν και ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη και την πολύ καλή συνεργασία. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις και για αυτή την, εργασία που ε, είχε αίσια πέραση. Περάσαμε ε, κάποια στιγμή για αρκετή συζήτηση με την πρωτοβουλία για το Youth Employment αλλά όπως είπαμε αν δούμε ότι μέσα στο 2018 δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια ένα, θα καταθέσουμε ένα διορθωτικό σχέδιο προπολογισμού και όπως είπε και ο Ρίτσαρντ θα υπάρξει μια αναθεώρηση για το δικαστήριο γιατί είναι αυτή η οποία, ε, το, αυτό το δικαστήριο το οποίο ε, φτιάχνει τη διαδικασία και εξετάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού και όπως βλέπουμε και στο διορθωτικό προπολογισμό 6 του 2017 το προϊόν των ε, προστήμων εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ε, είναι κατανοητό ότι χρειάζεται αυτή η, η, λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου. Αν ε, η διαδικασία κρατάει εξαιρετικά πολύ καιρό, αυτό αμφισβητεί ε, την ίδια τη λειτουργία της νοιάς αγοράς. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο χρειάζεται λοιπόν να έχει αυτά τα μέσα στη διάθεσή του για να μπορεί να διεκπαιρεώνει τις υποθέσεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Κύριε Καβίλιο, εσείς που ήσασταν παρούσα μονίμως, και διαρκώς ε, τρέχατε ανάμεσα στην αντιπροσωπεία του Συμβουλίου και, της, του Κοινοβουλίου. Μπορείτε να μας πείτε την, ποια είναι η εκτίμηση της Κομισιόν την επαύριο της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι εισηγητές, ε, αγαπητοί κύριοι, ε, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τη συμφωνία για τον προπολογισμό του 2018, στην οποία, την οποία καταφέραμε το Σάββατο στις πρώτες πρωινές ώρες μετά από εξουθενωτικές διαπραγματεύσεις. Όπως είπε ο κύριος Άσχορ, θα πρέπει όλα να τα θέσουμε μέσα σε μια προπτική. Έχουμε έναν προπολογισμό 160 δις ε, ακόμα και αν δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για όλα και κάποια λεπτομέρεια θα θέλαμε να, να έχει γίνει διαφορετικά, πάντως εν γέννη πιστεύω μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για αυτήν την εξαιρετική συμφωνία. Πολύ καλή συμφωνία. Η επίτευξη αυτής της συμφωνίας λοιπόν ήταν αρκετά δύσκολη παρά το γεγονός ότι φέτος οι θέσεις των δύο σκελών της Δημοσιονομικής Αρχής φαινόταν να είναι λιγότερο απομακρυσμένες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι θεσμοί είχαν κοινέ προλητικές προτεραιότητες, δηλαδή δημιουργία θέσεων απασχόλησης ασφάλεια, ε, ε, ήταν ωστόσο το ίδιο περίπλοκη όσο ανέκαθεν η διαδικασία και από την πλευρά της ε, Κομισιόν ε, έγιναν κάποιες σκληρές συζητήσεις και θέλω να τονίσω ότι και εμείς ήμασταν το ίδιο σκληροί και μετά τους δύο θεσμούς αλλά και δημιουργικοί γιατί καταφέραμε να συνδυάσουμε τις διάφορες θέσεις, να τις συμφιλιώσουμε με μεγάλες επιτυχίες και υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη διαπραγματευτική του ομάδα που έδειχνε την ίδια βούληση και αποφασιστικότητα ώστε να εξευρεθεί συμφωνία, ε, όπως την ίδια βούληση με εμά. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα σημεία που, που, που ε, ανέφεραν οι ομιλητές τους ή άλλως, αλλά Πιστεύω επίσης πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ικανοποιημένο με, ικανοποιημένο με το περιεχόμενο των αλλαγών που εισήχθησαν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα ο τίτλος 1α, σημαντικές αυξήσεις σε προγράμματα κλειδιά, επιτυχή προγράμματα, τα οποία είναι πολύ προσφυλή στο Κοινοβούλιο και η συμφωνία αυτή επετεύχθη με πλήρη σεβασμό στην ενδιάμεση <clears throat> αναθεώρηση που όπως ανέκαθεν λέμε δεν επηρεάζει τις αρμοδιότητες των σκελών της Δημοσιονομικής Αρχής στο πλαίσιο των διαδικασιών. Και όπως είπατε δικαίως κύριε Πρόεδρε ε, Αρτουή, και αυτές οι διαπραγματεύσεις φετινές το επιβεβαιώνουν αυτό. Ανέκαθ, ε, υπήρξε επίσης σημαντική αύξηση στον τίτλο 1β για την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που σηματοδοτεί τη σημασία που αποδίδουν οι τρεις θεσμοί στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Έχουμε και τη μονομερή δήλωση της ε, Επιτροπής ε, που μόλις αναφέρατε, ενίσχυση των ε, οργανισμών που ασχολούνται με την κρίση των προσφύγων, το προσφυγικό, Υπάρχουν και θέματα στο Global Europe που αφορούν την νότια γειτονία, την ανατολική γειτονία, όπου η πολιτική συμφωνία είναι απόλυτη ανάμεσα ε, στους θεσμούς ε, όπως είναι και το θέμα της χρηματοδότησης της Τουρκίας ε, και οι προτάσεις του Κοινοβουλίου για πιλωτικές προ... project και προπαρασκευαστικές δράσεις λήφθησαν υπόψη. Οπότε θα πρέπει αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη. Να συγχαρώ τη διαπραγματευτική ομάδα και κυρίως τον πρόεδρο Αρτουή φυσικά, τους εισηγητές μου Ρεσάν Ασουόρθο και Γκάγερ όχι μόνο σε σχέση με τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς, αλλά και με τον προϋπολογισμό του 18 είμαι πεπισμένη και προσβλέπω στη μεγάλη πλειοψηφία που πιστεύω πως θα έχει το Κοινοβούλιο ε, διακομματικά στην, ολο... στην ψηφοφορία στην Ολομέλη την άλλη εβδομάδα και ε, θα περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις του επόμενου Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε κυρία Καλβίνιο και ευχαριστώ για τη βοήθεια που μας προσφέρατε στη διάρκεια όλων αυτών των αναζητήσεων συμφωνίας. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές José Μανουέλ Fernández. Ε, θα, μιλάω, θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, να ευχαριστήσω ολόκληρη την διαπραγματευτική ομάδα, ε, τους ε, προέδρους, του, τους συζητητές, τον πρόεδρο Αρτουή που προσέφερε τη σοφία του και την εμπειρία του στο πώς να διευθύνει την ομάδα, στο πώς να διευθύνει τις διαπραγματεύσεις ώστε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο θεωρούμε επιτυχές και για το οποίο είμαστε όλοι περήφανοι. Και γι' αυτό και ε, ήθελα να το πω ρητά. Επίσης να ευχαριστήσω τον Γενικό Εισηγητή, τον Ζίκριτ Μουρεσάν, που έκανε εξαιρετική δουλειά, όπου ε, ε, συμμετείχαν όλες οι πολιτικές ομάδες. Έκανε εξαιρετική δουλειά επίσης. Να ευχαριστήσω τον Ρίτσαρτ Άσχουαρθ ο οποίος σε μια πάντοτε δύσκολη διαδικασία όπως είναι η διαπραγμάτευση για τα άλλα θεσμικά όργανα ε, πέτυχε το αποτέλεσμα. Για τους οργανισμούς επίσης ε, είναι δύσκολη υπόθεση και συγχαίρω τον συνάδελφο Γκάιερ ο οποίος κατάφερε να φέρει εις πέρας ε, για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες μας και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Όλους τους σκιώδες εισηγητές που συνέβαλαν σημαντικά ώστε αυτό το αποτέλεσμα να το πετύχουμε. Και Κάποιες ε, φορές δεν μιλάμε για το τι καταφέραμε πέρα από την πρόταση της Επιτροπής. Ξεχνάμε τις περικοπές που είχε κάνει το Συμβούλιο. 750, περικοπέ, 750 ε, ε, εκατομμύρια στο 1α είχε περικόψει το Συμβούλιο αρχικά. Εμείς αντιστρέψαμε αυτό το πράγμα και επιπλέον αυξήσαμε 250 ε, εκατομμύρια το προπολογισμό και ε, φέραμε νέο χρήμα σε κάποιους τίτλους που είναι η προτεραιότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήσαμε περισσότερη ανάπτυξη ε, και άρα έρευνα και ανάπτυξη, στήριξη στις εταιρείες και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλληλεγγύη εσωτερική και εξωτερική, ασφάλεια για τους πολίτες μας. Και αυτά όλα επετεύχθησαν χωρίς να ξεχνάμε ποτέ το, την πληγή αυτή τη, τη φοβερή της ανεργίας που δεν την ξεχνάμε ποτέ ε, πλήττει τους νέους ε, ενισχύσαμε την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων <clears throat> αυτό που φαινόταν μια δυνατότητα που ήταν η ενίσχυση με φρέσκο χρήμα προγραμμάτων σημαντικών όπως το ορίζοντας 2020 τελικά ε, βλέπουμε ότι καταφέραμε να εγκρίνουμε ότι η αναθεώρηση του PDP δεν θα προκαταβάλει τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε ετησίως για τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν είναι πάρα πολύ θετικό Ε, ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε τις ε, περικοπές που αντιστρέψαμε, τις περικοπές του Συμβουλίου και ένα, μια τελευταία λέξη για την Επιτροπή. Διαπιστώνω ότι σε αυτήν την διαπραγμάτευση διαπιστώνω την ισχύ, την πολιτική του Επιτρόπου, θέλω να πω. Και αυτό είναι πολύ καλό σημάδι και αυξάνει τις προσδοκίες που έχουμε για τα μελλοντικά μας θέματα. Ε, δουλεύουμε για πολύ σημαντικά θέμα, ε, και εμπιστευόμαστε την Κομισιόν και ελπίζουμε και ότι θα δείξει την ίδια δέσμευση τόσο η Κομισιόν όσο και το Κοινοβούλιο και κυρίως ο ίδιος ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Χωσέ Μανουέλα. Και τώρα θα δώσω το λόγο, όπως είπα, στους συντονιστές ή στους κοιόδης εισηγητές. Δανιέλε Βιώτη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να εκφράσω, ξεκινώντας τις ευχαριστίες μου προς τους εισηγητές ιδιαίτερα τον κύριο Μουρεσάν αλλά και τον κύριο Άσφορ, τον κύριο Γκάιερ και σε εσά βέβαια κύριε Πρόεδρε για τη δουλειά που κάνατε σε αυτές τις 16 ώρες διαπραγμάτευσης. που σας έφερε και σε αντιπαράθεση με το Συμβούλιο βεβαίως, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και ο Χουάν Φερνάνδες δεν θα τα ε, εκθέσω όλα τα επιχειρήματα. Θέλω να σημειώσω την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες προς τον εισηγητή και τον πρόεδρο για τα επιτεύγματα στον τίτλο 1α ιδιαίτερα. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς ε, να αρνηθεί την νίκη που καταγάγαμε σε αυτό το σημείο και πολιτική νίκη. 55 εκατομμύρια ευρώ αύξηση Δεν είναι μελιτέο ποσό. Είναι πολύ σημαντικό. Καθοριστική σημασία. Και ευχαριστώ τους εισηγητές και εσάς κύριε Πρόεδρε και για άλλα επιχειρήματα. Ξέρω βέβαια ότι κουραστήκατε ε, κοπιάσατε μάλλον πολύ να βρεθείτε ε, σε θέση να δώσετε επιχειρήματα απέναντι σε αυτό το να δύναμο κρίκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το Συμβούλιο. Το υπενθυμίσατε και εσείς. Ε, βρεθήκατε αντιμέτωποι με ένα Συμβούλιο, με έναν Υπουργό ουσιαστικά και από, την, ε, από τα άλλα κράτη ήταν όλοι αξιωματούχοι χωρίς ε, δυνατότητα και περιθώριο διαπραγμάτευσης έναντι των εντολών που είχαν από τις αρχές τους και τις κυβερνήσεις τους. Το δικό μας το περιθώριο και βέβαια και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερος, το δικό μας ε, επίσης το περιθώριο ήταν πολύ ε, ισχνό. Και έτσι πολλά από τα αιτήματα που είχε διατυπώσει το Κοινοβούλιο και είχαμε υποστηρίξει όλους αυτούς τους μήνες που έχτισε ο εισηγητής ε, κ. Μούρεσαν τον ε, προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Πολλές λοιπόν ε, από τις δικές μας διεκδικήσεις δεν ικανοποιήθηκαν, δεν βρήκαν απάντηση. είτε γιατί δεν δόθηκαν ε, απαντήσεις, είτε γιατί ο τρόπος με τον οποίο έγινε η συζήτηση από πλευράς του Συμβουλίου οδήγησε σε αυτό και με ξαφνιάζει, ε, δόθηκε έμφαση ιδιαίτερα σε αυτό που θα έπρεπε να είναι ένα αποτέλεσμα και όχι ένα σημείο κίνησης. Υπολογισμός δηλαδή των περιθωρίων. Από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση και όχι από τις ανάγκες και τις δεσμεύσεις που θα έπρεπε να τιμηθούν. Ε, και σε αυτό υπάρχει το πρόβλημα προς τον υπολογισμό των εμονικό θα έλεγα υπολογισμό των περιθωρίων από το Συμβούλιο. Επίσης και συμφωνώ με τον ε, κύριο Μουρεσάν, είχαμε την απόφαση για 80 εκατομμύρια μείων στον προϋπολογισμό το σχετικό με την Τουρκία στο κεφάλαιο 4 για τα προβλήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της, ε, του μη σεβασμού, της δημοκρατίας με όλα αυτά τα προβλήματα που γνωρίζει η χώρα. Λέμε αυτό και μετά βάζουμε στο αποθεματικό. Από φόβο η Τουρκία μας ζητήσει νέα ποσά το 2018 για το πρόβλημα το μεταναστευτικό των προσφύγων από τη Σύρια, τα ε, υπόλοιπα ποσά. Ε, αυτή ήταν η στάση των κρατών μελών, δηλαδή δεσμεύουμε χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, ε, που όμως το μεταξύ δεν έχουν καλύψει τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Και παρά τις προσπάθειες, το λέω, το επαναλαμβάνω, είμαι απολύτως πεπισμένος, παρά τις τεράστιες προσπάθειες και ευχαριστώ και πάλι του εισηγητή και όλους, όλης της ομάδας υπάρχουν στοιχεία που δεν μπορούν να μας ικανοποιήσουν. Δεν μπορούν να μας επιτρέπουν να πούμε ότι είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι. Ναι, μπορεί να έχουμε κάποια καλά ποσά σε άλλους τίτλους, τρία, τέσσερα, 5. Αλλά δεν, πήγαμε, δεν επισήλθαμε στη συζήτηση Τη ουσία. Δεν μπορέσαμε δηλαδή να εκθέσουμε του λόγου για του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμενε τόσο πολύ σε αυτού του τίτλου. Άρα αυτό που, εξασφαλίσαμε και σημειώνω ότι απέχουν πολύ τα ποσά από αυτά που έχει στήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το πρόβλημα λοιπόν πάνω από όλα είναι ότι δεν μπορέσαμε να πείσουμε το Συμβούλιο, δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε στο Συμβούλιο ποια είναι τα μελήματά μας, γιατί ζητάμε τα ποσά αυτά και χωρίς ε, να θέλω να καθυστερήσω τους λοιπούς συναδέλφους προχωρώ, στην, ε, προχωρώ για να ολοκληρώσω την ε, παρέμβασή μου. Πάλι στη μεθοδολογία κύριε Πρόεδρε, δύο ζητήματα. Πρώτον, ναι πολύ σύντομα. Με ενόχληση ιδιαίτερα η στάση του Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε τρία σημεία. Πρώτον, ότι στη συζήτηση για το 1Β εγγύηση για την νεολαία προσπάθησε προσπαθώ να βρω την κατάλληλη λέξη, προσπάθησε να αλλοιώσει τη συζήτηση δίνοντας ασφαλμένα στοιχεία σε σχέση με τη δυνατότητα απορρόφησης των ποσών από ορισμένα κράτη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε και να κάνουμε την επιχείρηση αλήθεια, δηλαδή να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Δεύτερο πρόβλημα για μένα, ε, μεθοδολογικό πάντα, είναι ότι στον τίτλο 4... Δεν έγινε σεβαστή η βούληση που είχε εκφραστεί και η συμφωνία για το ανθρωπιστικό ζήτημα που θα έπρεπε να καλύπτεται κατά 50% αν όχι κατά 100% για ορισμένες γραμμές του προϋπολογισμού. Η UNRWA για τους Παλαιστινίους που έχει αύξηση κατά 6 εκατομμύρια προς το παρόν μόνο στις ε, αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά 1,5 μόνο εκατομμύριο προβλέπεται για τις, αναλήψεις, για τις, ε, για τις πληρωμές. Επομένως δεν εξασφαλίζουμε ούτε κατά 50% τις ε, πληρωμές σχέση με τις αναλήψεις υποχρεώσεων και Τρίτο πρόβλημα που διαπιστώνω είναι ότι δεν τηρήθηκε καν η Συμφωνία Κυρίων που έχουμε εδώ και χρόνια και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως και στη σχέση με τα ε, όργανα μεταξύ τους. Κάποια πράγματα ναι, τα επιτύχαμε, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός ε, πλησιάζει αυτό που χρειαζόταν, όχι σε νούμερα μόνο, αλλά και σε σχέση με τις πολιτικές φιλοδοξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παρόλα αυτά ευχαριστώ τον εισηγητή, τους εισηγητές και τον Πρόεδρο γιατί ήταν ορατή η προσπάθεια και ο σωματικός ακόμη κόπος ε, στον οποίο αποδίθηκαν για τη δουλειά τους. Ο Πρόεδρος. Κύριε Τζότη, τουλάχιστον κάτι θα μπορούσε να σας ικανοποιήσει και, τον, ε, και εσάς βέβαια αλλά και το Γενικό Εισηγητή του 2019. ότι και το υπενθύμησε η κυρία Καλβινιό ότι η απόφαση για την εγγύηση των νέων ελήφθη χωρίς να χρειάζεται κάθε χρόνο να επανέρχεται το θέμα αυτό. Επομένως μπορούμε να το ορίσουμε και να το κλείσουμε με το midterm revision. Εσείς θα σας τάλλω στο Γενικό Σύγητης το 2019, οπότε θα έρθει η ώρα σας. Κύριος Κόλμελ, κύριος Βιώτη, πολύ σύντομα παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, θέλω να πω ακριβώς εδώ, πολύ γρήγορα, προσπαθώντας να μιλήσω πολύ γρήγορα, ξέχασα να σας πω αυτά στα οποία ήμουν ικανοποιημένο. Με συγχωρείτε, ο κύριος Κόλμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές, ε, τον κύριο Μουρεσάν, τον κύριο Άσχορτ και τον κύριο Κάιερ και να ευχαριστήσω όχι μόνο να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ και τον Πρόεδρο γιατί θεωρώ ότι το αποτέλεσμα είναι πραγματικά μαξιμαλιστικό. Είναι ακριβώς αυτό που αναγνωρίζει την πραγματικότητα και νομίζω ότι πρέπει από την πλευρά μου να κάνω μια αποτίμηση. Δεν βλέπω τόσο αυτή την αντι... αντιπαράθεση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Εμείς ως Κοινοβούλιο έχουμε πολλές ε, ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε με τα λεφτά και είναι και τα, τα κράτη-μέλη αυτά που δίνουν τα λεφτά. Οπότε καταλαβαίνετε ε, τελείως διαφορετικά σκέφτονται αυτοί από εμάς στο Κοινοβούλιο. Ε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και νομίζω ότι υπάρχουν και πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Έχουμε καλά αποτελέσματα. Στη γενική γραμμή να πω ότι ε, έχω ικανοποίηση, όμως ε, δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε μια άλλη κατεύθυνση σε αυτόν τον προϋπολογισμό και υπόθηκε ήδη Υπάρχουν ε, πολλές ε, πολιτικές ε, καταστάσεις που δεν έχουν αναγνωριστεί. Μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό που μπορέσαμε να δεσμευτούμε για την ανεργία των νέων και αυτό είναι σωστό και είναι καλό όταν υπάρχουν σωστά project να παίρνουν χρήματα. Όμως αυτό τελικά παρακάμπτει τα τα αίτια, τα πραγματικά. Κοιτάμε μόνο τα συμπτώματα. Εκεί που είναι υψηλή η ανεργία των νέων πρέπει να πατάξουμε τα αίτια. Και αν θέλουμε αυτά να τα αντιμετωπίσουμε θα ήταν πιο πολύ σημαντικό ε, να δώσουμε χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση παρά ε, στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των συμπτωμάτων. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές ε, γραμμές που εδώ και δεκαετίες παραμένουν στο ίδιο και ε, τελικά ε, ο τρόπος που έχουν καταναμηθεί τα κονδύλια εκεί ε, πλέον είναι παροχημένος. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα και νομίζω ότι τελικά δεν ήταν και τόσο μεγάλη η επιτυχία. Υπάρχουν βέβαια πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Το είπαμε ήδη σήμερα. Είπαμε ότι θα θέλαμε από ε, κοινού να κάνουμε κάποια πράγματα στο θέμα της άμυνας. Νομίζω ότι και πάλι δίνουμε τη λάθος κατεύθυνση. Ε, κανείς δεν λέει πώς θα πρέπει να είναι αυτή η κοινή άμυνα ε, γιατί φαίνεται ότι είναι δύσκολο να μιλάμε για τόσα μεγάλα ποσά τελικά που πρέπει να χρηματοδοτήσουν ε, τα κράτη-μέλη, όπως ας πούμε στον τομέα του ασύλου. Ε, εκεί τι πρέπει να πετύχουμε. Αυτό πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε, με ποια μέσα, με ποια μέτρα και πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν έναν τέτοιο προϋπολογισμό και δυστυχώς αυτό δεν πραγματοποιείται. Ευχαριστούμε τον κύριο Κόλμερ, ο κύριο Τάραντ. Έχετε το λόγο, κύριε Τάραντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρεις παρατηρήσεις έχω, για να μην επαναλάβω και τα συγχαρητήρια και όλα όσα ήδη υπόθηκαν και σωστά υπόθηκαν. Παρατήρησα για πρώτη φορά ε, στη ζωή μου ότι υπήρξε μεγάλη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, αυτή τη συμφωνίας της συνδιαλλαγή ως ένα μεγάλο γεγονός ε, και πραγματικά πρέπει να είναι μεγάλο το επίτευγμα για να γίνεται αυτό. Δεύτερον, αυτό συγχαίρομαι που δεν μπορούσα να λάβω μέρος στις διαπραγματεύσεις γιατί συνήθως όταν είμαι εκεί δεν είναι εύκολο κανείς να φτάσει σε συμβιβασμό και τρίτον ανησυχώ λίγο με αυτή την επερχόμενη ψηφοφορία στις Βρυξέλλες γιατί αν ε, ε, θυμάστε μπορεί να υπάρξει και πρόβλημα νομικό. Είμαστε νομικά υποχρεωμένοι αυτά να τα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. Αν αποφασίσουμε λοιπόν ε, να πάμε το θέμα στο Στρασβούργο, ίσως μπορούμε να αποφύγουμε δαπάνες δικονομικές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, σας αναγνωρίζουμε τόσα λέτε. Ο κύριος Χριστοφόρου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει, ε, δεν υπάρχει πραγματικά καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται σήμερα για μια μεγάλη επιτυχία της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Και αυτή η επιτυχία πιστώνεται στον πρωταγωνιστή αρχικά, στον κύριο Σίκρι Μουρεσάν, στο Προεδρείο της Επιτροπής και σε όλους τους αγαπητούς συναδέλφους που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί είναι μεγάλη επιτυχία να κατορθώνει σε αυτή την περίοδο να πετυχαίνει αυξήσει για το Horizon, για το Erasmus, για το κόσμο, για του νέου ανθρώπου, για του νέου αγρότε, για του άνεργου νέου, για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, την ανάπτυξη, την έρευνα, προσδίδεται μια άλλη κοινωνική διάσταση στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνεται το μήνυμα ότι αυτή η Επιτροπή έχει τεράστιε ανεπτυγμένε ευαισθησίε για την κοινωνία αλλά και για την ανάπτυξη και την οικονομία. Δεν μπορώ να μην θεωρήσω σημαντική επιτυχία το ότι κατορθώσαμε να περικοπούν κονδύλια 105 εκατομμυρίων στην Τουρκία για να σταλεί ένα μήνυμα. Όμω η πάγια διαχρονική θέση και άποψή μου είναι ότι δεν μπορούν χώρε οι οποίε παραβιάζουν συλλήβδη και αντιστρατεύονται τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, που δεν σέβονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πολλές φορές προσέβαλαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν έστω έναν ευρώ χρηματοδότηση. Η Τουρκία δεν μπορεί να λαμβάνει καμία χρηματοδότηση και καμία άλλη χώρα που συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Δεν είναι μόνο για την Τουρκία. Όμω δεν μπορεί ταυτόχρονα μια χώρα να συνεχίζει να κατέχει χώρα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθημερινά να προκαλεί, να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και εμείς να ζητούμε έστω να χρηματοδοτείται, έστω κατελάχιστο η Τουρκία. Πιστεύω ότι αν ρωτήσουμε σήμερα τους Ευρωπαίους φορολογούμενους πολίτες εάν πρέπει η Τουρκία να παίρνει έστω έναν σεν από τα ευρωπαϊκά ταμεία η απάντηση θα είναι καθολική όχι. Και σίγουρα οι δικοί μου Ευρωπαίοι πολίτε, οι Κύπροι πολίτε, με τίποτα δεν δέχονται να συνεχίσει να χρηματοδοτείται αυτή η χώρα έστω και με ένα ευρώ. Όμω, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να εκφράσω τι ευχαριστίε μου προ την Επιτροπή και στου αγαπητού συναδέλφου και στον αγαπητό εισηγητή, τον Σίκριφ, γιατί για μια ακόμη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε ευαισθησία για ένα μείζονο σημασία ανθρωπιστικό ζήτημα που είναι το θέμα των αγνωμένων η διερεύνηση τη τύχη των αγνωμένων στην Κύπρο εδώ και 43 χρόνια, όπου δίνονται επιπρόσθετα 2 εκατομμύρια ευρώ. Που και εδώ θέλω να σα ενημερώσω ότι και για αυτό το ανθρωπιστικό θέμα η Τουρκία συνεχίζει να προβάλλει εμπόδια να μην ανοίγει κλειστού χώρου και να μην ανοίγει τα αρχεία του στρατού για να διερευνηθεί η τύχη των αγνωμένων. Θεωρώ σήμερα ότι πραγματικά δικαιούμεθα να περηφανευόμεθα ότι υπήρξε μια σημαντική επιτυχία της Επιτροπής Προϋπολογισμού για τον προϋπολογισμό του 2018 και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε το μήνυμα ότι το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το μέλλον και την προοπτική αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πέρασε μέσα από τόσα προβλήματα και από τόσε δυσκολίε. Για μια ακόμη φορά συγχαίρω του αγαπητού συναδέλφου που πρωταγωνίστησαν και του ευχαριστώ για την ανταπόκριση και στα δικά μα αιτήματα. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ε, και ευχαριστώ όλη την ομάδα των εισηγητών, ε, καθέναν από τους συναδέλφους. Ε, θέλω να χαιρετήσω την εξαιρετική τους δουλειά και την αντοχή διότι ήταν πολλοί οι μήνες που δουλέψαμε ε, για αυτό τον προϋπολογισμό του 2018. Αν μου το επιτρέπετε, γιατί ο κύριος Φερνάντες δικαίως μίλησε για το επίπεδο των απαιτήσεων και ακριβώς περί αυτού πρόκειται σε ποιο επίπεδο βάζουμε τις απαιτήσει μας για τον προϋπολογισμό του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έλεγα και κρίμα που κάποιοι έχουν φύγει. Πάντως αυτό το επίπεδο των απαιτήσεων δεν είναι το τίμημα των απαιτήσεων του Κοινοβουλίου αλλά συχνά είναι προϊόν ε, των ετοιμάτων του Συμβουλίου για νέες πολιτικές που σωρεύονται. Αυτή η διατήρηση λοιπόν αυτού του επίπεδου απαιτήσεων ε, μας οδηγεί να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι το ίδιο ε, ε, για την Επιτροπή του Προπολογισμού για όλους είναι αυτό αξιοσέβαστο και δεν θα πρέπει να, πώς να το πω, να χαλάσει την ατμόσφαιρα ούτε και να διαβρώσει την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Απλά να διαπιστώσουμε ότι δεν είμαστε αναγκαστικά όλοι στο ίδιο επίπεδο απέτησης. Γιατί η πολιτική, η συμβολική και η ψηφιακή ακόμα ε, νίκη θεωρώ Ε, αφορά μόνο το ένα α και για τα υπόλοιπα κάτι ψίχουλα καταφέραμε. Και το είπατε και δικαίως κύριε Πρόεδρε ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ότι ε, ποιες ήταν, οι περιορισμοί και για τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις και αν όμως δεν είχαμε κάνει τα λάθη που είχαμε κάνει σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις θα μπορούσαμε σίγουρα να πάμε και να καλύψουμε τα λάθη των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Αυτό κατά τη γνώμη μου. Πέρα λοιπόν από αυτή την πολιτική νίκη που είναι αξιοθαύμαστη, κατά τα λοιπά, εγώ, εμένα μου μένει μια πικρία. Και, και το είπα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Υπάρχει μια μορφή ε, ανηλικρίνειας από πλευράς του Συμβουλίου, την οποία δεν ανέχομαι. Ο Ντανιέλ Εβιώτη το είπε πριν από λίγο, ότι στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν από περιθώρια τα οποία δεν ήταν αποδεκτά, όλοι γνωρίζουμε πως δεν ήταν διαπραγμάτευση για τα περιθώρια, αλλά ότι ήταν διαπραγμάτευση επί τη ουσία για την διευκόλυνση για την Τουρκία και το Συμβούλιο δεν θέλησε να το βάλει στο, στη βιτρίνα της διαπραγμάτευσής του. Κυρία Καλβίλιο, πριν από λίγο είπατε πως ε, είστε ικανοποιημένοι και περιμένατε με χαρά τις επόμενες διαπραγματεύσεις του Νοεμβρίου 2018 για τον προπολογισμό του 2019 ε, εγώ δεν, το, δεν χαίρομαι και τόσο. Θα σας πω, πω τι εγώ ε, αισθάνθηκα και πάλι δεν είμαι εισηγήτρια, δούλεψα πολύ λιγότερο από τους ίδιους τους εισηγητές. Να σας πω ότι όταν μας δίνουν ε, τις τροπολογίες σε τρεις μέρες πριν τη διαπραγμάτευση και όταν μας καλούν να κλειδαμπαρωθούμε στο Συμβούλιο για μια νύχτα μέχρι ότου τελικά να εγκρίνουμε πεθαμένη στην πείνα γιατί με εκείνα τα τρία μικροσκοπικά σαντουιτσάκια κλειδαμπαρωμένοι στο συμβούλιο ήμασταν μέχρι να πούμε ναι. Εγώ παρενόχληση. Ναι, όχι, όμοιρος αισθάνθηκα, όμοιρος. Πολύ μου κακοφάνηκε. Ναι, αλλά ο Γκάγερ είχε κρατήσει όμοιρο το διορθωτικό προπολογισμό του 2017. Ναι η ομοιρία ενός προπολογισμού δεν είναι η ομοιρία ανθρώπων. Εγώ ειλικρινά την επόμενη φορά δεν ξέρω πώς, αλλά δεν μπορεί να γίνει έτσι. Όχι. Μας ταπείνωσαν, το κοινοβούλιο το ταπείνωσαν. Συγγνώμη, τα λέω λίγο όπως τα σκέφτομαι. Εγώ είχα την αίσθηση της ταπείνωσης στη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης. Δεν λέω, και το είπε και ο Λαντανιέλε Βιώτη, δεν μιλώ για τη στάση του Συμβουλίου που μας στέλνει έναν κατακαημένο ε, υπάλληλο του Υπουργείου, ενώ όλοι οι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρελάβουν στο Γκέτεμποργκ για ένα κοινωνικό πυλώνα που δεν έχει καμία νομική αξία, ούτε καν ε, δημοσιονομική αξία, αλλά εκεί πάνε κάνουν τους, ε, τους ωραίους και παρελάβουν ψωροπερήφανοι αλλά εκεί που είναι η ουσία για τα δημοσιονομικά ούτε μισός υπουργό δεν ήρθε. Ε, μα δεν είναι αυτή η κατάσταση. Εγώ αισθάνομαι ότι ε, δεν με σέβονται και εφόσον δεν με σέβονται δεν σέβονται ούτε τον Ευρωπαίο πολίτη. Πραγματικά μεγάλη πικρία κρατώ από αυτή τη διαπραγμάτευση. Συν ότι ήμουνα με άδειο ε, στο μάχη. Λοιπόν, συγγνώμη, τα λέω λίγο έξω από τα δόντια, αλλά αυτά είναι δικά μου και τα λέω. Ευχαριστώ που μοιράζεσαι μαζί μας αυτές τις, ε, ε, τα συναισθήματα. Κύριο κύριος Ρούμπιχ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι ικανοποιημένο από τις ε, διαπραγματεύσεις γιατί προχώρησαν όπως πάντα. Ίσως αν ήταν παρόντες υπουργοί να ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι εύκολο ίσω για του υπουργού να είναι παρόντε για ένα πολύ μικρό προπολογισμό. Εξού αυτό για το επόμενο έτο μα επιτρέπει να μείνουμε περισσότερο και να μιλήσουμε για την συνθήκη της Λισαβόνας, για το 1% του ΑΕΠ που είναι, λιγότερο, που είναι κάτω από το 1% ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και για, για το δεύτερο και τρίτο δεκαδικό ψηφίο για το οποίο φτάσαμε μέχρι τις 3 το πρωί και τις 4 το πρωί για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Πρόκληση λοιπόν. Εγώ από αυτό, όλο αυτό καταλήγω στο εξής συμπέρασμα. Για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε για το 1.24. Στον ορίζοντα 2020 το Συμβούλιο έδειξε μια κάποια ευελιξία και σε αυτό ευχαριστώ και τον Επίτροπο αλλά και την ομάδα του. Μπορέσαμε να φτάσουμε στα 110 εκατομμύρια. Ήταν σωστή η έμφαση που δόθηκε και οι προτεραιότητες και νομίζω ότι αυτό θα δώσει θα έχει και τον αντίκτυπό του στον πολίτη. Θα το δει ο πολίτη και θα το αναγνωρίσει, άλλωστε και τα μέσα μαζική ενημέρωση θα ενημερώσουν. Αν και συνήθω δεν το πράττουν, αν δεν δουν κάπου σκάνδαλο όπου γίνεται σωστά η δουλειά, λησμονούν να ενημερώσουν του πολίτε. Μετά είδαμε, περιμέναμε πρωινό, πρωινό δεν ήρθε να προσφερθεί. Μπορέσαμε να κλείσουμε τη δουλειά εγκαίρως ε, για την αναθεώρηση για τα κτίρια βγήκανε τα 5 εκατομμύρια σε σχέση με την ε, συμφωνία κυρίων που είχαμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή έγινε σεβαστή καλή εξέλιξη Νομίζω ότι δείξαμε πνεύμα και ανοχή και κατανόηση. Φυσικά υπάρχει ανάγκη και για αμοιβαιότητα στις στάσεις μας το ένα όργανο απέναντι στον άλλον για να έχουμε μια καλή συνεργασία. Και χαίρομαι που δεν χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι τρίτη το πρωί της τρέχουσας εβδομάδας για να σκάσει η διαπραγμάτευση για να αποτύχει δηλαδή. Κερδίσαμε πολλά, κάναμε μεγάλες οικονομίες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω... Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις εδώ στο Κοινοβούλιο, οπότε την οικονομία την κάναμε εμείς. Επίσης θα ήταν καλό να ξέρουμε ότι πρέπει να πιέζουμε να γίνεται η διαπραγμάτευση στη συνδιαλλαγή και στον τριμερή διάλογο εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί εμείς έχουμε τότε το πάνω χέρι, εμείς ορίζουμε το πρωτόκολλο, τη σειρά, ε, τη διάρκεια και αν ε, είναι δυνατόν, ε, εάν δεν είναι δυνατόν να πιέσουμε για περισσότερο, τότε θα πρέπει πότε μία και πότε, πότε από εδώ και πότε από εκεί να γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πάντως κύριε Αρτουή, κύριε Πρόεδρε, ιδιαιτέρως για τη διαχείριση όλου αυτού του έργου και για τη μεγάλη σας επιτυχία. Φυσικά και θα μπορούσαν ακόμα καλύτερα να γίνουν, αυτό το ξέρουμε όλοι, αλλά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Merci. Donc, euh, Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Παρακαλώ τον εισηγητή Ζήξιτ να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι από την πλευρά μου. Καλός ο προϋπολογισμός. Εκεί είναι τα αποτελέσματα 105 για το 1α, 160 για το β, 35 για το 4. Έχουμε τους οργανισμούς στον τομέα της άμυνας πιο ισχυρο, ισχυρούς. Ίσως δεν έχουμε αρκετά σάντουιτς, αλλά ίσως να έχουμε του χρόνου περισσότερα. Το ελπίζω. Ρίτσαρτ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, Πρόεδρε Γιάννης. Ούτε εσύ. Όχι. Ωραία, ευχαριστώ συνάδελφοι. Νομίζω ότι πρέπει τώρα να αποφανθούμε. Στο Στρασβούργο. δεν βλέπει κανείς κάποιο ε, μειονέκτημα. Πρέπει μέσα σε δέκα μέρες ε, ε, μετά τη συμφωνία να αποφανθούμε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δόθηκε λοιπόν στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής ε, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα ε, του συνδιαλλαγής ε, και θα προσαρτηθεί στο πλήρες κείμενο του προϋπολογισμού για το 2018-29 Νοεμβρίου λοιπόν στις Βρυξέλλες είναι η, είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια και 30 η ψηφοφορία. Η Επιτροπή θα εκφραστεί για τα τέσσερα πακέτα τα οποία αφορούν στη διαπραγμάτευση και θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Το μέσο ε, ευελιξίας, ε, το Ταμείο Αλληλεγγύης ε, και ο Δημοσιονομικός διορθωτικός προϋπολογισμός 6 για το 2017. Όλα αυτά θα είναι στο πακέτο. Ελπίζω λοιπόν ότι με την ψηφοφορία μας θα μπορέσουμε να θέσουμε την Ευρώπη εν κινήσει και όχι στο περιθώριο. Και τώρα ο κύριος ε, Ζαμπάλα για την ετήσια έκθεση με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η κυρία Ρουμπιάλ. Ευχαριστώ θα τα πω κι εγώ σύντομα. Ναι, νομίζω ότι είναι εύκολο να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Όπως έλεγα θα είμαι σύντομη γιατί ε, έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο σε αυτή τη συζήτηση και μάλιστα ε, δεν πίστευα πως ε, θα κάνουμε μεγάλη συζήτηση εδώ, ε, γιατί το ε, κάναμε την ημέρα της παρουσίασης της έκθεσης. Να δούμε μόνο τις τροπολογίες που λάβαμε, ήταν 21 τον αριθμό. Είναι αλήθεια ότι πολλές από αυτές και στην πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων είναι παρόμοιες μεταξύ τους και στην ίδια γραμμή με αυτά που είχα ήδη εγώ αναφέρει στη διάρκεια της συζήτησης της έκθεσης και είναι πολύ συμπληρωματικά θα μπορέσουμε, πιστεύω, να βρούμε συμφωνία για κάθε, ένα από, κάθε μία από τις τροπολογίες και κάθε ε, η δική μου ε, ένδειξη για την ψηφοφορία θα είναι θετική. Θα πρέπει να μειώσουμε ε, να δούμε και ποιες είναι οι φιλοδοξίες μας σε σχέση με αυτή την έκθεση. Να αναγνωρίσουμε λοιπόν ε, τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να, κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο, τη διαφάνεια και ούτω καθεξής. Εγώ θέλεις αυτά να τα αναδείξω, αλλά... Να αναγνωρίσουμε λοιπόν τη δουλειά που κάνουν, αλλά πιστεύω πως θα πρέπει και να συνεχίσουμε πιέζοντας ώστε να συνεχίσουν να βελτιώνονται όπως λέει και η παρουσίαση, ώστε να μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για συστήματα ελέγχου, λογοδοσίας και διαφάνειας. Άρα λοιπόν πιστεύω πως αυτή είναι η φιλόδοξη μας πρόταση, να συγχαρώ και τους συναδέλφους, αλλά και να συνεχίσουμε όπως είπα να απαιτούμε ε, να δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν πως ε, θα χρειαστεί να υποβάλουμε και κάποιες συμβιβαστικές γιατί όπως έλεγα οι περισσότερες παράγραφοι προχωρούν προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι τροπολογίες που μπορούν να προσθεθούν άμεσα. Ε, παράγραφος 8 και παράγραφος 11 έχω παρόμοιες τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να δουλέψουμε για μια τροπολογία, κυρίως την 11 γιατί όταν δουλεύουμε για μια τέτοια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είχαμε φτάσει ε, στη σε συμφωνία στο FC2 και άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε και να προσθέσουμε τις τροπολογίες που έχουμε. Κάποια σχόλια συγκεκριμένα, γιατί έλαβα διάφορες τροπολογίες από διάφορες πολιτικές ομάδες που ζήτησαν, θέλησαν μάλλον να τονίσουν και να καταδείξουν κάποιες υποθέσεις, κάποιες περιπτώσεις, κάποια project που χρηματοδότησε η ΕΤΕΠ που ήταν αμφίβολα ή, εν πάση περιπτώσει, όχι και πολύ ορθά, ορθά. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει ανά περίπτωση όντως να τονίζουμε και να βάζουμε ονοματεπώνυμο στα συγκεκριμένα, στα προβλήματα σε μια τέτοια γενική έκθεση αξιολόγησης των δραστηριοτήτων. Γιατί έτσι θα είναι ένας τρόπος ο καθένας να καταδείξει το project που δεν λειτουργήσε και να ξέρουμε ότι αυτό είναι και ο στόχος της έκθεσης. Ε, θέλουμε να στραφούμε στο μέρον και άρα ο έλεγχος των δραστηριοτήτων το, το, της ΕΤΕΠ γίνεται από την Επιτροπή Έλεγχου του Προϋπολογισμού. Ε, ε, ο εξονυχιστικός τώρα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα για την ώρα. Νομίζω δεν έχω μεγάλη στήριξη εδώ, αλλά δεν θα τα παρατήσω. Προσπαθώ να βρω η στήριξη τις επόμενες μέρες. Έχει να κάνει με την αποζημίωση της εγγύησης και με την τιμή. Την τιμολόγηση, το pricing, είναι μάλιστα ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί και στη διάρκεια της συζήτησης για την έκθεση FC2. Το διαπραγματευτήκαμε το Συμβούλιο με την Επιτροπή και με την ΕΤΕΠ επίση. Για μένα είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα και πιστεύω ότι θα μπορέσουν οι πολιτικές ομάδες, θα τους να στηρίξω αυτή την παράγραφο. Γιατί όσο, τόσο η αποζημίωση της εγγύ... η κατάθεση εγγύησης όσο και η το είναι πράγματα τα οποία μπορούν να τροποποιηθούν, να βελτιωθούν σε ορισμένους τομείς, σε ορισμένες ε, είδη επιχειρήσεων και μπορεί να ταιριάξουν καλύτερα σε ορισμένες χώρες γιατί η κατάσταση τραπεζική δεν είναι η ίδια στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία, στη Γαλλία ή στη Ρουμανία. Άρα λοιπόν απαιτούμε από την ΕΤΕΠ να προσαρμόσει και να, και να χρησιμοποιήσει καλύτερα αυτά τα εργαλεία ώστε να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις σε όσες περισσότερες χώρες γίνεται στην Ένωση. Και η τιμολόγηση επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ώστε να αναγνωριστεί τη θέμενη αξία, το θετικό στοιχείο κάθε project ε, ένα είδος βραβή, βράβευσης σε πάση περιπτώσει ε, αυτά τα project που δεν είναι τραπεζικά μόνο, είναι ενδιαφέροντα οικονομικά από οικονομικής άποψης και από κοινωνικής άποψης και θα είναι δηλαδή ενδιαφέρον να χρηματοδοτηθούν, να προωθηθούν εν περιπτώσει γιατί επιδιώκουν καλύτερα τους στόχους, στηρούν καλύτερα τα κριτήρια και ούτω καθεξής. Να χρησιμοποιηθεί λοιπόν αυτή η τιμολόγηση ως ένας τρόπος προσέλκυσης αυτών των ε, project. Ε, αλλά εδώ υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις στις απόψεις ε, και δεν ξέρω. Ε, θα προσπαθήσω εγώ να υποβάλω μια πρόταση. Ένα τελευταίο σχόλιο. Μια-δύο παράγραφοι σε σχέση με την εξωτερική εντολή τη ε, ΤΕΠ. Επειδή είμαστε σε διαπραγματεύσει και μάλιστα έχουμε αρχίσει νέο γύρο διαπραγματεύσεων και αύριο έχουμε τριμερή, θα ήθελα να αφήσω αυτή την ενημέρωση αυτή τη παραγράφου μέχρι το τέλο, ώστε να δούμε τι στήριξη θα έχουμε, ελπίζουμε, και αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία, μακάρι, για την εξωτερική εντολή της ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, Εντέρ, για αυτή την διαφωτιστική σου έκθεση και για ε, αυτή την ε, ΤΕΠ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον ε, θρησκειώδη ηγετή που σας, μας συνοδεύει, τον κύριο Αλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίως Θέλω να υπογραμμίσω ξεκινώντας την ε, ποιότητα της δουλειάς σου και κάποιες από τις προτάσεις. Ο ρόλος της τράπεζας βεβαίως είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Αυτό είναι ουσιοδέστατο στοιχείο. Η επίλυση των ε, τρέχουσών πολιτικών προκλήσεων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως δεν πρέπει να είναι η μόνη ή η κύρια ε, προσέγγιση. Πρέπει να μιλούμε για κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Πρέπει να περιλάβουμε το λειτουργικό πρόγραμμα 2017-2018 που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο. Προσανατολισμοί, επιδόσεις, κύριες δραστηριότητες δηλαδή για τα επόμενα τρία χρόνια. Η τράπεζα ετοιμάζει το προσεχές λειτουργικό σχέδιο 2018-2020, τριετές πάλι. Οι άλλες προτάσεις στις ε, προσφυγές ή παράπονα. Έχουμε να κάνουμε με μια προσέγγιση της ΕΤΕΠ σε σχέση με, συνεργα... με μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες ή κράτη και την πολιτική εναντί αυτών. Μια αναθεώρηση δηλαδή των ε, σχετικών επιλογών σε σχέση με αυτές τις τράπεζες. Ε, αντίστοιχη προσέγγιση είχαμε και στο παρελθόν. Λογοδοσία. Η ΤΕΠ έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση της πολιτικής για τους καταγγέλλοντες με, ένα, με μια επιχείρηση μέσω προσδιορισμού οροσίμων έχουμε προχωρήσει ήδη για να δώσουμε έναν απολογισμό αυτών των δραστηριοτήτων. Επίσης δραστηριότητες της ΣΤΕΠ σε σχέση και με την λογοδοσία προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να αποδίδουν μόνο για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που διαχειρίζεται ο όμιλος της ΣΤΕΠ ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι δεν αναμειγνύουμε με εντολές ε, άλλου τύπου που αναλαμβάνει η ΤΕΠ. Ευχαριστώ κυρία Λύη. Κύριος Χωσέ Μανώλη Φερνάντες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Secret Μουρεσάν. Ο κύριος Μουρισάν χρειάστηκε να αποχωρήσει γιατί έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Τον εκπροσωπώ λοιπόν. Ευχαριστώ ιδιαίτερο τη συνάδελφο ε, για τη δουλειά της, εξαιρετική δουλειά. Και βέβαια η αριστεία, όπως θα λέγει η κυρία Τωμά, εξαρτάται από τις φιλοδοξίες μας. Θα, αν ήμουν η κυρία Τωμά θα έλεγα εξαιρετική έκθεση, αλλά, αλλά και θα προσέθετα κι άλλα μετά, αλλά τη βγάζω την παρένθεση αυτή, διότι ομιλώ εκ μέρους του κυρίου Μουρεσάν ο οποίος ε, συμφωνεί με τα περισσότερα στοιχεία της έκθεσης και τις ε, τροπολογίες. Βεβαίως η Επιτροπή συμβάλλει από πλευρά της έτσι ώστε όλα τα κράτη να έχουν και την απαραίτητη mm. ικανότητα πρόσβασης ε, τεχνογνωσία πρόσβαση στα εργαλεία που διαθέτει η ΤΕΠ και αυτή η ΕΤΕΠ θα πρέπει να προσφέρει και την τεχνική υποστήριξη έτσι ώστε να περιορίζονται οι γεωγραφικές αποκλήσεις και να αποκλείονται στο μέγιστο όπως ορίζεται και στην τροπολογία 14. Στην 121 μιλούμε για την συνεργασία μεταξύ εθνικών τραπεζών ανάπτυξης που πρέπει να έχουν αυτή την ε, συνεργατική σχέση με τα διαφορετικά ταμεία και τα μέσα επενδύσεων. Και εδώ ιδιαίτερα τονίζουμε αυτά τα μέσα που έχει διαθέσει τη ΣΥΕΤΕΠ ε, προκειμένου να επιτευχθούν ε, οι στόχοι. Υποστηρίζουμε το iCredit Standing και το τριπλό α, υψηλή δηλαδή πιστοποίηση πιστοληπτικής ικανότητας, ε, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί και ε, επικίνδυνα ή επίφοβα έργα η ΕΤΕΠ όχι μόνο με στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα και σε γειτονικέ χώρε που έχουν ανάγκη να υποστηρίξουν τη δημοκρατία του, να δίνει τα μέσα για τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει. Δεν πρέπει να λησμονούμε ασφαλώ τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει που είναι ιδιαίτερα σημαντικέ για την οικονομία μα. Σα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντε, κύριο Σάνι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και πολύ σύντομα Στο το είπε και η συγκήτρια, θα είναι λίγα τα σημεία συμβασμού γιατί λίγο πολύ έχουν ικανοποιηθεί τα σημεία. Δύο ερωτηματικά μόνο, σημαντικά για μένα. Πρώτα απ' όλα, και το συζητήσαμε και σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018 ε, για την Τουρκία. Όχι μόνο δεν παίρνει τα κονδύλια, όχι μόνο παίρνει τα, κονδύλια του προενταξιακού μέσου Τουρκία, αλλά και πάρα πολλά κονδύλια μέσω της χρηματοδότησης της ΕΤΕΠ, περισσότερα από κάθε άλλο κράτος. Πολλά, ε, από πολλά τουλάχιστον κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που ε, μαθαίνω από την απόφαση που ελήφθη Ε, από τη διαπραγμάτευση αυτή για τον προϋπολογισμό είναι ότι όταν υπάρχουν κάποιες ε, ε, όταν υπάρχει η βούληση πολιτική μπορούμε με ό,τι και να συμβαίνει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και άρα μπορούμε να πιέσουμε την, την ΕΤΕΠ στηριζόμενοι και στις αποφάσεις του Γενικού Προϋπολογισμού σε σχέση με τις πιστώσεις που διατίθενται σε αυτήν τη χώρα για να ακολουθούν οι πιστώσεις αυτές κριτήρια όχι μόνο και όχι αυστηρά, όχι μόνο και εξαντλητικά οικονομικά, αλλά και κριτήρια δημοκρατίας, κράτους δικαίου κτλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε έναν επαναπροσδιορισμό αυτής της, της ε, αιρεσιμότητας των ε, κονδυλίων που αφορούν την Τουρκία για να ξαναγυρίσουν τα λεφτά στην Ένωση. Επίσης, πρόσβαση στα δεδομένα η ΕΤΕΠ είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία οικονομικά εργαλεία στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωση, το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δημόσιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του κόσμου και μπορεί να φέρει, ε, να δώσει απαντήσεις, να εξασφαλίσει ε, εξελίξεις θετικές και πολύ σημαντικές ως προς την οικονομία συγκεκριμένων κρατών. Έτσι λοιπόν εμείς ως συνομοθέτες, η Επιτροπή, το ελεγκτικό συνέδριο είναι απαραίτητο να έχουμε πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό όγκο δεδομένων για τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΤΕΠ. Πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε πάντα στο παρελθόν. Έχουμε μια τελευταία έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που επισημαίνει την ε, ε, ανεπάρκεια των δεδομένων που διατίθενται από την ΕΤΕΠ και γι' αυτό θα πρέπει να καλέσουμε την ΕΤΕΠ να ενισχύσει στο πεδίο της επικοινωνίας τα στοιχεία που διαθέτει και κυρίω στο βαθμό που ε, προσφέρει ε, στις, στα θεσμικά όργανα, τα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφορίες αυτές. Για να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να αξιολογούμε καλύτερα τις δραστηριότητες του χρηματοπιστωτικού αυτού ιδρύματος και ε, να βεβαιωνόμαστε ότι οι στόχοι που έχουμε εμείς ορίσει για το έργο της ΕΤΕΠ υλοποιούνται και κατά τρόπο μάλιστα μετρήσιμο αντικειμενικά δεδομένου ότι ε, και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία. Κυρία Μάλετιτς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση, όπως και τους σκιώδεις για τη συνεισφορά τους. Ως εισηγήτρια για την γνωμεδότηση της Επιτροπής Ρέτζη θα ήθελα να τονίσω ότι μας εξέπληξε λίγο το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε και εγώ δεν μπόρεσα να βρω συγκεκριμένες ε, πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ΕΤΕΠ σε σχέση με την πολιτική συνοχής παρόλο που κοιτώντας το άρθρο 308 της συνθήκης βλέπουμε πως ε, ορίζεται ότι η ΕΤΕΠ πρέπει να ε, υποστηρίζει τις, ε, τις περιοχές αιστέρηση και να υποστηρίζει και την ευθυγράμμιση της αγοράς. Επίσης τονίζεται ότι η ΕΤΕΠ πρέπει να μειώνει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Και τέλος, δεν υπάρχει ειδικό κεφάλαιο στην έκθεση της ΕΤΕΠ για αυτές τις δραστηριότητες και για το πώς ακριβώς υποστηρίζεται η μείωση των ανισοτήτων. Παρόλο που, κοιτώντας τις δραστηριότητες που είναι υποχρεωμένοι να εκτελέσουν, καταλαβαίνουμε ότι έχουν φτάσει στις επιχειρησιακές δυνατότητές τους στα σε επίπεδο κρατών μελών, υπάρχει και η συγχρηματοδότηση. Θα ήταν εύκολο λοιπόν να υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο και μια ειδική έκθεση για αυτά. Ελπίζω όλα αυτά να μπουν και στην τελική έκθεση. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να αναλύουμε με λεπτομέρεια σε ποια χώρα δίνεται οικονομική υποστήριξη Τελικά, όταν το κοιτάξαμε, είδαμε πως σε πέντε κράτη-μέλη δίνουν πάνω από το 50% των συνολικών δανείων. Άρα, όλα πάνε στα πέντε πιο ε, πλούσια κράτη. Και αυτό το λέει στη... δεν είναι αυτό που λέει η συνθήκη. Αν δούμε επίσης τη θεματική συγκέντρωση θα δείτε ε, ακριβώς πώς αυτή σχετίζεται με τις μεταφορές, την ενέργεια, τη βιομηχανία που είναι καλό. Επίσης ε, πάνω από τα μισά ε, δάνεια κατευθύνεται προς αυτές τις θεματικές προτεραιότητες, όμως θεωρώ ότι πρέπει να πάμε περισσότερο προς την καινοτομία, την ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υποστηρίζουν την καλύτερη μεγέθυνση και ανάπτυξη στα κράτη-μέλη. Π.χ η επιστήμη και η σχέση της επιστήμης με την πραγματική οικονομία η οποία υποστηρίζεται με νέες ιδέες. Ήθελα απλώς να τονίσω όλα αυτά, να τα έχετε στο μυαλό σας, ότι χρειάζεται να περιλαμβάνετε στην έκθεση και η μείωση των ανισοτήτων. Ευχαριστώ. Eh Ευχαριστώ. Όσοι θέλησαν να μιλήσουν μετά την εισηγήτρια το έκαναν. Τώρα πρέπει να μιλήσει η ΕΤΕΠ μέσω της κυρίας ε, Αντώνη που είναι η Γενική, Διευθύν, Γενική Γραμματέας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να συμβάλλω κι εγώ στο διάλογο σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ για το 2016. Με χαρά μου Ακούω τους επένους που λαμβάνει η ΕΤΕΠ για τις δραστηριότητες της, όμως θα ήθελα να τονίσω ένα πράγμα. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω ότι στην ουσία αυτό που κάνουμε εμείς είναι να ε, υποστηρίζουμε τις επενδύσεις. Είμαστε ο επενδυτικός βραχίωνας. Ο όγκος λοιπόν των επενδύσεων που εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε έχοντας αναλύσει με το μακροοικονομικό μοντέλο της ε, κοινή υπηρεσία έρευνα τη Κομισιόν, ε, τι δυνατότητέ μα, ε, ε, είναι αυτό που θα σας παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Με βάση λοιπόν αυτά που έχουμε και την οικονομική έρευνα, να πω ότι η ΕΤΕΠ είναι ο επενδυτικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει τις πολιτικές σχετικά με τις επενδύσεις. Για την διαφάνεια έχουμε αυξήσει τις προσπάθειές μας να μεγιστοποιήσουμε τη διαφάνεια και τις πληροφορίες που δίνουμε για τα διάφορα project. Και όχι μόνο τα project που έχουν να κάνουν το εργαλείο στρατηγικών επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, αλλά και με οποιαδήποτε άλλο εργαλείο, με όποιο project είναι διαθέσιμο. Ε, τα βλέπετε όλα στην ιστοσελίδα μας. Δημοσιεύουμε επίσης τις εκθέσεις του Συμβουλίου και τα πρακτικά και στην, πρακτική, πολιτική της διαφάνειας να πω ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε οποιοδήποτε έγγραφο ζητούν οι ενδιαφερόμενοι. Θα το ξέρετε. Κατανοώ βέβαια ότι οι πληροφορίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμε. Ως τώρα έχουμε τον, τη συνοχή. Η συνοχή είναι το 20% των συνολικών μας στόχων. Όπως ξέρετε έχουμε άλλους στόχους δημόσιας πολιτικής, καινοτομία, περιβάλλον, υποδομές και μικρομεσές και μετά έχουμε τους οριζόντιους που είναι η κλιματική δράση και η συνοχή. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των στόχων πολιτικών που καλύπτουμε. Επίσης, ε, να έλθω τώρα στο θέμα των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Όπως ξέρετε, έχουμε μια πολιτική που είναι στα σπάργανα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να την ε, εξετάσουμε, την ε, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ακριβώς. Επίσης για τα άλλα θεσμικά όργανα να πω ότι έχουμε αυξήσει τα μοντέλα συνεργασίας κυρίως λόγω ε, της υποστήριξης από την εγγύηση. Έχουμε πολλά μοντέλα συνεργασίας και χθες είχαμε μια συνάντηση με την Κομισιόν και διερευνήσαμε ακριβώς ε, πώς ε, θα κάνουμε το διάλογο με τα εθνικά ε, Ινστιτούτα Προώθησης, τα National Promotion Institutions, για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά είναι και πολύ σημαντικά να έχουμε και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα τα επιτρέπει. Γι' αυτό ο συνδυασμός των κονδυλίων ΕΣΥΦ και είναι σημαντικός θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερη και πιο συνεκτική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων θεσμικών ε, οργάνων. Τώρα να έρθω στις αμοιβέ ε, για την ε, εγγύηση. Η ΕΤΕΠ είναι φυσικά τράπεζα και έχουμε και τα προϊόντα τα οποία τιμολογούνται βάσει των αγορών του κινδύνου. Την αγορά εργασία κοιτάμε δηλαδή για την τιμολόγησή μας. Κάποιε φορέ είναι δύσκολο. Τέλο πάντων, πώ να το πω, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε η τιμολόγηση να μην είναι ο κινητήριος μοχλός, να είναι άλλοι παραγοντές οι οποίοι θα καθιστούν άριστο ένα project. Οι δυνατότητες που θα δίνονται στις εταιρείες και τους ενδιάμεσους χρηματοδότες, όλα δηλαδή αυτά τα άλλα στοιχεία ε, που διέπουν ένα project για να μην έχουμε στρέβλωση της αγοράς που δεν θέλουμε φυσικά. Και για την ε, πολιτική για τις μη συμμορφούμενες δικαιοδοσίες και την φορολογία να πω ότι συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την καθοδήγηση αυτής. Επίσης, περιμένουμε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που θα πρέπει να δημοσιευθούν το Δεκέμβρη και πρέπει ε, να προσαρμόσουμε και την πολιτική μας για τις μη συμμορφούμενες δικαιοδοσίες NCJ πώληση. Τον, ε, τον Δεκέμβρη θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά προς το παρόν. Χαίρομαι ιδιαίτερα ε, και το επαναλαμβάνω πρόεδρε που ο διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είναι πολύ σημαντικός για μας. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Μαθαίνουμε πολλά και είμαστε και χαρούμενοι που μπορούμε να σας στείλουμε και ένα follow-up report όπως έγινε και πέρυσι. Θέλουμε, ότι είναι σημαντικό. Θέλουμε να γίνεται αυτό γιατί είναι σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και για τα όσα μας είπατε και δεν αμφιβάλλω ότι όλα όσα υπόθηκαν το πρωί από τους συναδέλφους θα τα λάβετε υπόψη σας στην ΕΤΕΠ. Αυτά. Θέλετε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτή την ανταλλαγή. Κυρία Έντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, πολύ σύντομα. Γιατί τα περισσότερα σχόλια τα έχουμε ήδη συζητήσει και οι τροπολογίες που μας εξήγησαν τόσο οι φιλελεύθεροι όσο και το ΕΛΚ θα ληφθούν υπόψη γιατί συμφωνούν με τη γραμμή εργασίας που είχαμε ήδη χαράξει. Είναι κρίμα που έφυγε ο κύριος Τζάνι γιατί αναφέρθηκε στην Τουρκία και νομίζω πως είναι σημαντικό να τον ενημερώσω. Α, εδώ είστε πίσω μου. Ωραία, τέλεια για το θέμα της Τουρκίας, γιατί μάλιστα έχει μεγάλη σχέση με τις συζητήσεις που κάνουμε με την εξωτερική ε, εντολή της ΕΤΕΠ. Βλέπουμε ε, ότι η Επιτροπή, η ΕΤΕΠ και το Συμβούλιο και εμείς έχουμε την ίδια άποψη ότι πρέπει να μειώσουμε την έκθεση της ΕΤΕΠ στην Τουρκία και να ε, εκμεταλλευτούμε αυτά τα κονδύλια που θα απελευθερωθούν για να τα διανύμουμε σε άλλους τομείς που θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητα στο Κοινοβούλιο. Αυτό, αυτό ωστόσο δεν έχουμε μπορέσει να το συζητήσουμε με το Συμβούλιο ακόμα. Ε, πάντως, ε, εν γέννη φαίνεται να υπάρχει αυτή η γραμμή μείωση των, της στήριξης της ΕΤΕΠ ε, προς τα project της Τουρκίας. Σε σχέση με την γνωμοδότηση της ΡΕΤΖΙ και της ΕΚΟΝ, αναφερόμαστε σε, αναφέρονται συγκεκριμένα θέματα. Μόλις χτες εγκρίθηκαν, οπότε δεν έχω ε, ε, σχόλια ε, για να μπορέσουμε να τα λάβουμε υπόψη ακόμα. Ωστόσο, να ευχαριστήσω για τα σχόλια που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή πολιτική και την αλήθεια ότι η ΕΤΕΠ ε, δεν έχει ακόμα απαντήσει. Τουλάχιστον να μείνει ε, γραπτά οι φόβοι και οι απορίες που έχουμε. Και αυτό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την πολιτική διαφάνειας και πρόσβαση στην ενημέρωση και η ΤΕΠ κάνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το τομέα. Ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε να πετούμε να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το δρόμο. Γιατί κάποιες φορές είναι δύσκολο, κυρίως στο Κοινοβούλιο, να βρούμε τέτοιες πληροφορίες. Ε, είναι αλήθεια ότι... Ε, ε, εμείς ερχόμαστε σε επαφή άμεσα με την τράπεζα για να μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες. Αν ψάξουμε όμως στο ίντερνετ δεν υπάρχουν πάντα αυτές τις πληροφορίες. Τελευταίο μου σχόλιο για το pricing. Ε, καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι τράπεζα και δουλεύει με βάση την αγορά. Ωστόσο δεν μπορούμε να ξεχνάμε, αλλά δεν είναι και, και τράπεζα κερδοσκοπική και δεν είναι μια τυχαία ε, τυχαία τράπεζα γιατί η εγγύηση στις ε, είναι ένας δημόσιος προϋπολογισμός. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά της ΕΤΕΠ σε σχέση με άλλες ε, τράπεζες. Άρα λοιπόν όχι μόνο η τιμή είναι σημαντική, η τιμή θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο τα, έχει να κάνει με αυτά τα project και η τεχνική αρρωγή είναι θεμελιώδης, είναι ένα από τα βασικά πλονεκτήματα που προσφέρει η ΕΤΕΠ στους ε, προσθέτες αυτής της τράπεζας, ωστόσο δεν μπορούμε να στρεβλώσουμε την αγορά. Καταλαβαίνω ότι τηρώντας αυτές τις, τις προϋποθέσεις θα πρέπει και η τιμή να είναι ελκυστική για τα διάφορα project. Να, να ε, σεβόμαστε τις συνθήκες που ισχύουν λοιπόν στην αγορά και να στηρίζουμε τα project όχι μόνο μέσα από την τιμή αλλά και μέσω της προστιθέμενης αξίας που αντιπροσωπεύει η, η ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα γίνει τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Και τώρα θα κάνουμε, θα δούμε πού βρίσκεται ο τριμερής για την απλοποίηση του χρηματοπιστικού κανονισμού. Απλοποίηση. Ελπίζω να μην είναι ψευδής διαφήμιση αυτή η λέξη. Ο Ashworth είναι ε, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, μου φαίνεται ότι είναι υπεραισιόδοξος όρο, όρος, τελικά. Δέκα είναι οι τριμερείς διάλογοι που έχουμε πίσω μας και μας λείπουν 20 σελίδες για να ολοκληρώσουμε την πρώτη αναγνώση των κανονισμών. Άρα υπάρχει κάποιο φως. Καλό αυτό γιατί είναι δεδηλωμένη η βούληση όλων των πλευρών ώστε μέχρι το τέλος της Εστονικής Προεδρίας τον Δεκέμβριο να έχουμε τελειώσει αυτό το έργο. Αφενός μεν γιατί θα είναι πρακτικά αδύνατον η Βουλγαρική Προεδρία που ακολουθεί να πάρει πάνω της όλο το έργο, να προετοιμαστεί και να το συνεχίσει. Θα είναι τελείως παράλογο να περιμένει κανείς ότι θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια δουλειά. Και επιπλέον διότι οι Επιτροπές Γεωργίας και Περιφερειακής Πολιτικής έχουν ολοκληρώσει το δικό τους μέρος της δουλειάς για το πακέτα Omnibus. Σήμερα μάλιστα η Γεωργική έκλεισε τη συμφωνία της, τις προτάσεις της και είναι απαραίτητο να έχουμε τις προτάσεις αυτές έτοιμες για την 1η Ιανουαρίου. Τούτου λεχθέντος. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα για τα 74 άρθρα που πρέπει να ξαναδούμε στο μέλλον. και θα έχουμε και άλλους ε, τριμπέρις διαλόγους. Από την τελευταία φορά λοιπόν που σας ενημέρωσα εδώ συζητήσαμε και εξετάσαμε και επαληθεύσαμε διαδικασίες απαλλαγής και δημοσιονομικού ελέγχου και κυρίως το ανέφερε ο Πρόεδρος ε, το Κοινοβούλιο θέλει προ... πρωταρχικά να απλοποιήσει και δευτερευόντως να επιταχύνει τις διαδικασίες. Θέλουμε δηλαδή το χρονοδιάγραμμα καταρχάς για τις απαλλαγές να είναι πιο πιεστικό, δηλαδή ε, ε, το αργότερο στο έτος νήσιν ένα να έχει ολοκληρωθεί η απαλλαγή, σε αυτό συμφωνούμε. Επίσης, έχουμε μια σειρά από θέματα στη διαδικασία του δημοσιολογικού ελέγχου, όπου πάλι δεν έχουμε καταλήξει συμφωνία προς το παρόν και θα ήθελα να υπενθυμίσω στους κοιόδης, αγαπητέ Πρόεδρε. Δευτέρα βράδυ συνεδρίαση. Είναι απαραίτητο να είναι παρόντες, είναι απαραίτητο να γίνουν αυτές οι συζητήσεις μεταξύ μας πριν περάσουμε στον τριμερή διάλογο. Όχι την ώρα που είναι να εξελίξει ο τριμερής διάλογος. Αυτά και ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά. Θα θέλω να τόσο φόρο τιμής στην προσήλωσή σας, το τιτάνιο έργο σας, το συναρπαστικό αυτό δημιούργημά σας και τα επιτεύγματα στο πλαίσιο των προσεχών πολιτών δημοσιονομικών προοπτικών πάντως οπωσδήποτε πρέπει και ο δημοσιονομικός κανονισμός να αναθεωρηθεί γιατί από αυτά που ακούω μέρα με τη μέρα έχει γίνει κατάσταση αφόρητη. Είναι σε ένα βαθμό αποτελεσματικός αυτός ο κανονισμός. Γιατί όμως, γιατί ο δικαιούχος παρετείται από τη διεκδίκηση των κονδυλίων με όλους τους ελέγχους, τους εξπός, τους εξάντε, τους κατά τη διάρκεια, με όλο αυτό το κλίμα της απόλυτης δυσπιστίας έναντι των δικαιούχων που δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως έχει, διότι ε, αναιρεί κάθε αξιοπιστία της Ευρώπης στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη και δίνω το λόγο του του λεχθέντος στον αγαπητό κύριο Μάνκα που είναι σκιώδης συγητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να, καταρχάς να συγχαρώ σύντομα τον εισηγητή. Έχω λάβει μέρος σε έναν από τους τριμερείς διαλόγους. Όταν ένας μέσα σε δύο μήνες, ε, ένας άνθρωπος πρέπει να λάβει μέρος σε δέκα τριμερείς διαλόγους, ε, πραγματικά είναι μεγάλο εγχείρημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν, ήταν ε, πολύ καλή η προετοιμασία, πηγαίνουν άριστα οι διαπραγματεύσεις και έτσι θα μπορέσουμε το, του χρόνου να προχωρήσουμε με αυτό το ψήφισμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν και να ζητήσω ε, να αντέξετε μέχρι το τέλος γιατί πραγματικά οι δικαιούχοι περιμένουν από μας τα χρήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκράσλερ. Ε, δυστυχώς ε, δεν μπορεί να είναι εδώ. Παρόλο που είναι πάντοτε διαθέσιμη και έχει και μια εμπειρογνωμοσύνη που τη θαυμάζουμε και βασιζόμαστε πολύ πάνω της. Ε, είναι αυτή που θα απλοποιήσει τα πράγματα, όμως δεν μπορεί γιατί η Επιτροπή Άγκρη δεν μπορεί να απλοποιήσει τον ε, κανονισμό και αυτά μέσα στα μέσα του ε, πολιτές δημοσιονομικού πλαισίου του χρόνου λοιπόν για το επόμενο πολιετές Ζητήθηκε να γίνει κάτι τέτοιο, όμως δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και υπάρχει μια επίγουσα ανάγκη για πραγματική απλοποίηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο θα εμπνέεται από την λογική της εμπιστοσύνης και όχι της δυσπιστίας. Αφόσον τα είπαμε αυτά και εφόσον κανείς άλλο εκτό ε, από τον κύριο Μάνκα δεν ζητά το λόγο και κανείς άλλος δεν θέλει να προσθέσει κάτι, να δώσω το λόγο στον κύριο Άσχουερθ. Ελπίζω ότι μέχρι τα τέλη του χρόνου θα ολοκληρώσουμε το Omnibus Agri θα είναι έτοιμο για να κατατεθεί στην Ολομέλεια πριν τα τέλη του έτους. Διότι υπήρχε κάποια αμφιβολία σχετικά με αυτό οι διατάξεις ε, στο Omnibus ε, θα μπορούν να μπουν σε ισχύ ε, στην αρχή του επόμενου έτους για τον τομέα της γεωργίας. Ωραία. Πάμε τώρα σε μια συζήτηση πρώτης προτεραιότητας. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που η Ευρώπη υποστηρίζει στην Αφρική και να υποδεχτώ τους προσκεκλημένους, τους, κύρους, τους κυρίους Κόρμπενσε και Ρομπέρτο Ρουντόλφτη από την ε, ε, Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ και τον εκπρόσωπο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Ήδη τον ακούσαμε σε μία ανταλλαγή απόψεων το Μάρτι με τις Επιτροπές ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ. Έχουμε την ε, Αφρικανική Εβδομάδα. Είχαμε την Αφρικανική Εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την πέμπτη εβδομάδα που θα γίνει στο Αμπιτζάν 29 και 30 Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος Ταγιάννη σήμερα το απόγευμα θα κάνει και ε, κάποια ανοιχτή εκδήλωση το απόγευμα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τις επιτροπές ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ. Ε, που έχουν προσκεκληθεί. Ε, η πρόεδρος Μακέιβαν. δεν ξέρω αν είναι εδώ. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα γίνει ως εξής. Πρώτος, ο κύριος Ντόνσκ θα μας πει ποια είναι τα εργαλεία χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Μετά θα πάμε στον κύριο Ριντόλφη, ο οποίος θα μας δείξει πώς ε, οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ε, αϊφόρο ανάπτυξη ε, συμπληρώνουν και αλληλεπιδρούν με τα υφιστάμενα εργαλεία και θα δούμε και τους διάφορους οικονομικούς ε, παράγοντες που δρούν στην Αφρική. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κόντονς, ε, που είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να ξεπεράσετε τα 12 λεπτά στην παρέμβασή σας για τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην Αφρική. Ευχαριστώ. Υπόσχομαι να είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα, Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο καταρχάς που ετοιμάσε αυτήν την συνεδρίαση που είναι πολύ ε, χρήσιμη. Ξεκινάμε λοιπόν για την Αμπιτζάν για να προετοιμάσουμε βέβαια και την προσεχή Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικανικής Ένωσης πολύ σημαντική διότι θεωρούμε και το βλέπουμε και από τις συζητήσεις ε, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια νέα συνειδητοποίηση, ενισχυμένη συνειδητοποίηση στην Ευρώπη της σημασίας της Αφρικής. Και έχουμε αρχίσει λοιπόν να εξετάζουμε νέους τρόπους για να βλέπουμε την ε, Ήπειρο την Αφρικανική. Και αυτό που συμβαίνει στην Αφρική θέλουμε να μην μένει στην Αφρική. Ξέρουμε ότι οτιδήποτε συμβαίνει στην Αφρικανική Ήπειρο άμεσα επηρεάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα αυτό που βλέπουμε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη γεωγραφικά ήπειρο με τεράστιες προκλήσεις δημογραφική έκρηξη αλλά και μεγάλες ευκαιρίες και ως προς το δημογραφικό μέρισμα και ως προς την οικονομική ανάπτυξη, τεράστιο δυναμικό σε πολλούς τομείς, γεωργία καταρχάς, δυναμικό προστασία σε παραδείγματι δημιουργία, παραγωγή ε, ε, ενέργειας. Είναι ένα δυναμικό τεράστιο και το να βοηθήσουμε τους Αφρικανούς εταίρους μας να αναπτύξουν, να ε, αποδεσμεύσουν, να απελευθερώσουν αυτό το δυναμικό θα έχει τεράστια σημασία. Έχουμε να κάνουμε με πληθυσμό νεαρό, ιδιαίτερα νεαρό. Μέχρι το 2050 θα έχει διπλασιαστεί και άρα θα είναι ο πιο νέος ζωτικός ε, του κόσμου μέχρι τότε. Άρα λοιπόν σημειώνεται μια αλλαγή προτεραιοτήτων σε Πεντευρωπαϊκή Ένωση, που αντικατοπτρίζει πιστεύω και την αλλαγή προτεραιοτήτων ε, στην ε, ε, στο παγκόσμιο θεματολόγιο για την ανάπτυξη έχουμε περάσει από μία θεώρηση του 2015 που αναφερόταν στους στόχους της χιλιετίας, της χιλιετίας. Τώρα έχουμε το θεματολόγιο του 2030 με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που βέβαια κλειδώνει πάνω στο θεματολόγιο για την Αφρική. Το θέμα αυτή της συνόδου είναι οι οικονομικές δεσμεύσεις μας εναντί της Αφρικής Και θέλω να ξεκινήσω με ένα χαρακτηριστικό στοιχείο ότι εμείς στην Αφρικανική Ήπειρο είμαστε παρόντες και δεσμευόμαστε με τρία διαφορετικά εργαλεία. Τρία γεωγραφικού χαρακτήρα, το ενδέκατο ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το DCI ιδιαίτερα όσο αφορά την Νότια Αφρική, το DCI είναι πολύ ενεργό και βέβαια έχουμε και το εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία. Έχουμε επίσης τα θεματικά πρόγραμμα, προγράμματα του DCI, έχουμε το Παναφρικανικό, Έχουμε το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Δημοκρατίας Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, το Εργαλείο για τη Συμβολή στη Σταθερότητα και την Ειρήνη και το EDF μέσα στο ΑΚΕ που πάλι έχει γεωγραφικό προσδιορισμό την Αφρική και κυρίως, όχι αποκλειστικά όμως, το, ευρωπαϊκό, το Αφρικανικό Εργαλείο για την Ειρήνη ε, ιδιαίτερης σημασίας και δυνατοτήτων που μας επιτρέπει να δραστηριοποιούμαστε σε τομείς που δεν θα είχαμε τη δυνατότητα υπό τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό να αναλάβουμε δράση. Όλα αυτά λοιπόν ε, σημαίνουν ένα σημαντικό ποσό για το 2014-2020 αναμένεται συνολικά να δεσμευθούν 31 δισεκατομμύρια ευρώ για την Αφρική. Χρήματα που ανήκουν στη στην διαχείριση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν συμπληρωθούν αυτά και με τις συμβολές φορές των κρατών μελών, το ποσό γίνεται εντυπωσιακά υψηλό. Για το 2015 Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη συνολικά 21,4 δις είχαν δέσμευση για την αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική. Αυτό, αυτή λοιπόν η χρηματοδοτική προσέγγιση και προσήλωση δέσμευση για την Αφρική που μας καθιστά πρώτο χορηγό ε, θα πρέπει να έχει και ένα αντίκρισιμο πολιτικό. Είμαστε βεβαίως ο μόνο ένα εταίρο και τη ορισμένοι άλλοι και δι, οι Κινέζοι έχουν ήδη ξεκινήσει μια σαφή ε, λήψη θέσεων έναντι της Αφρικής αλλά έχουμε πολύ μεγάλες εμπορικές συναλλαγές το 3% των εισαγωγών της Αφρικής και το, 60%, το 40% των εξαγωγών της Αφρικής είναι σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε το νούμερο ένα για τις, ε, πρώτες, για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και πρώτη σε ποσά ε, αποστελόμενα με εμβάσματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρική. Έχουμε λοιπόν 21 ε, δις εμβάσματα από τους ε, ομογενείς, τους Αφρικανούς που είναι στην Ευρώπη. Και Συμπληρώνω για να πω ότι έχουμε μια σειρά από εργαλεία στη θέση μα για τη δραστηριότητα και τι δεσμεύσει μα στην Αφρική. Το έχετε συστήσει, φαντάζομαι, και με τον Επίτροπο Μίμητσα. σω στο μέλλον, λοιπόν, θα ήταν σκόπιμο να εξετάσουμε αυτό το περίπλοκο νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα και να διαρωτηθούμε αν υπάρχει δυνατότητα για πραγματικέ προσπάθειε που θα μα επιτρέψουν να ε, συντονίσουμε κάπως αυτά τα δημοσιονομικά μέσα για να τα απλοποιήσουμε, να τα διευκολύνουμε και να καταργήσουμε τους ε, τεχνητούς φραγμούς μεταξύ τους, έτσι ώστε να δώσουμε ουσιαστικές απαντήσεις στους, ε, στις ανάγκες της Αφρικανικής Ήπειρου, κύριας προτεραιότητας της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο σχόλιο σχετικό με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσουμε αυτή τη δέσμευση, δηλαδή αν υπάρχει μετατόπιση σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους εργασίας, τη χρηματοδότηση των project, με προς, μάλλον προς νέα, όχι νέα, αλλά με όλο και μεγαλύτερη έμφαση πλέον, νέα μέσα και νέους τρόπους. Ε, καταρχάς, ε, δημοσιονομική υποστήριξη, ενίσχυση που επιτρέπει και πολιτικό αντίκρισμα στις επενδύσεις και καλύτερη απόδοση των επενδύσεων, πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Αφενός, αφετέρου δε, και αυτό θα σας το εξηγήσω Ρομπέρτο καλύτερα, εγγυήσεις και ανάμιξη κονδυλίων μέσω του νέου EIP οι εγγυήσεις. Και έτσι έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα αλλά και καλύτερη χρήση των κονδυλίων της αναπτυξιακής βοήθειας για να αποδεσμεύσουμε, να απελευθερώσουμε άλλα κονδύλια που είναι χρήσιμα συνδυαστικά και δεδομένων των τεράστιων προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Αφρική πρέπει έτσι να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η κατάλληλη λύση, να χρησιμοποιούμε την αναπτυξιακή μας βοήθεια έτσι ώστε από πλευρά της αυτή να μοχλεύει, να αποδεσμεύει άλλα ποσά, σημαντικά ποσά είτε από δημόσιε, είτε από ιδιωτικέ επενδύσεις και αν μου επιτρέπετε θα σταματήσω εδώ. Αυτό ήταν εισαγωγικό σε σχέση με τη συζήτηση. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Μιλήσατε. Σας είχα δώσει 12 λεπτά και εσείς μιλήσατε για 8 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε συντόμως και πριν να δώσω το λόγο στην κύριο Ρινόλφη, νομίζω θα ήταν καλό οι συνάδελφοι που θέλουν να ε, κάνουν παρατηρήσεις για τα όσα μας είπατε να πάρουν το λόγο τώρα. Θα ήθελε κάποιο, ο κύριο Ντεπχέ. Κύριε Ντεπχέ μου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είμαι ειδικό στα όσα μα είπατε, Όμω. Αλλά μου κίνησαν το ενδιαφέρον δύο νούμερα που αναφέρατε και τα ποσά είναι συγκρίσιμα. Ότι είπατε για κάποια περίοδο η παρέμβαση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει το 21,5 δις και ότι αυτά αν κατάλαβα καλά αντιστοιχούν στα όσα στέλνουν οι Αφρικανοί που έχουν φύγει από την Αφρική ε, στους δικούς του στην, Ήπειρο, στην ίδια χρονική περίοδο. Αν λοιπόν διπλασιάζαμε τον αριθμό των Αφρικανών που έρχονται να δουλέψουν εδώ, αντί να έχουμε όλη αυτή τη γραφειοκρατία, <laughs> τι θα άλλαζε. Voilà, c'est la première question, monsieur. Εδώ η πρώτη ερώτηση, Κόλμπερν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα ε, παρουσία. Ήταν σύντομη αλλά είχε περιεχόμενο να είμαι σύντομος ε, στις σκέψεις μου. Μιλήσαμε για δυνατότητες απλούστευσης και ακούσαμε πόσο περίπλοκο είναι αυτό το ε, μόρφωμα ε, των διαφόρων ενδιαφερομένων για την Αφρική. Ε, έτσι θεωρώ λοιπόν ότι από τη μία μεν είναι περίπλοκο αλλά από την άλλη είναι πολύ σημαντικό παρά το γεγονός ότι ούτως ή άλλως πρέπει να δώσουμε χρήματα ε, για ανθρώπους που είναι σε ανάγκη να κοιτάμε και τι πετυχαίνουμε με αυτά τα χρήματα δηλαδή η παροχή ε, βοήθειας, ενίσχυσης να συνδέεται με την κατάσταση ειδικά ε, βάσει των όσων βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Την τεράστια μεταναστευτική κρίση η οποία συνδέεται άμεσα με την Αφρική. Για να είμαι ειλικρινής πρέπει να βλέπουμε όλες τις δυνατότητες αλλά και ακριβώς ε, και τις ε, άλλες διαστάσεις που έχουν να κάνουν με το πού απευθύνονται οι στόχοι και πώς ε, αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες. Θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει? Αν μου το επιτρέπετε να μιλήσω κι εγώ. Γιατί η Αφρική για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Οι δημογράφοι μας ανακοινώνουν ότι ο πληθυσμός της Αφρικής θα πάει πολύ πάνω από τα 800 εκατομμύρια, ε, ε, θα φτάσει στο 1 δις στα επόμενα χρόνια. Αυτό φυσικά δημιουργεί μια άλλη κλίμακα. Και οι πολλοί είναι οι Αφρικανοί οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ε, μια τεράστια και κρίσιμη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε δείξει τα διάφορα μέσα, αλλά δεν υπάρχουν τελικά υπερβολικά πολλά μέσα και ελάχιστες πιστώσεις για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας. Πραγματικά ο κίνδυνος είναι μίζων και κρίσιμος. 4-5 21,5 ε, είναι τα δημόσια κονδύλια τα οποία δίνονται ε, για αυτό το θέμα, δις, και η Αφρικανική Διασπορά ε, θα θέλει και αυτή το αντίστοιχο. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με την εργασία, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με τη δημόσια ενίσχυση που δίνεται. Εγώ σκέφτομαι τη Γαλλία, την χώρα στην οποία εκλέχθηκα. Υπάρχει το δημόσιο χρέος ε, υπάρχουν ε, χρήματα που ε, υπάρχει δημόσια βοήθεια που δίνεται στους Αφρικανούς που ζουν στη Γαλλία και όλοι πρέπει τελικά να αναρωτηθούμε τι κάνει το κάθε κράτος μέλος, τι κάνει η Ευρώπη. Δεν έχει έρθει πια η στιγμή, κύριοι διευθυντές, να ζητήσουμε από τα κράτη-έθνη να συνεργαστούν λίγο περισσότερο, να έχουν μια καλύτερη συνεργασία με τις παλιές τους απικίες και που κάποιες φορές ε, είναι λίγο προβληματική. Αυτά είναι τα θέματα που ήθελα να θίξω, κύριοι διευθυντέ. Ταυτόχρονα πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ζήτημα αυτό είναι μέγιστης σημασίας. Και δεν είναι απλώς μια γειτονιά. Ε, πρέπει να θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα στην πηγή τους. Να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλάνο για την Αφρική, να έχουμε μια εταιρική σχέση με τις αφρικανικές αρχές για να αναλαμβάνουν και αυτές τις ευθύνες τους, έτσι ώστε να φρενάρουν λίγο τις μεταναστευτικές ροές. Γιατί μιλάμε για οικονομικούς μετανάστες. Και ε, φυσικά Πολλά κράτη-μέλη ε, θα πρέπει, της πολλά μέλη, κράτη της Αφρικής θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να επιστρέψουν οι άνθρωποι αυτοί στη χώρα τους τελικά. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω για όσα μας παρουσιάσατε, αυτά που είπατε, τις αναλύσεις. Ε. Φαίνεται ότι ε, ο πληθυσμός ε, θα αυξηθεί ε, υπερβολικά στην Αφρική μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Τόσοι άνθρωποι θα ζουν στην ανέχεια, εκατοντάδες εκατομμύρια μετανάστες θα έρθουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιες δεσμεύσεις. Πρώτον, ως προς την εκπαίδευση των νέων, για να μπορέσουμε να πατάξουμε τη φτώχεια. Α, δεύτερον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην Αφρική και γι' αυτό χρειαζόμαστε και αναλύσεις που θα λένε τι μπορεί αυτό να κοστίσει. Μπορεί και σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις, όπως είπα, να κάνουμε έναν διάλογο για την αναπτυξιακή βοήθεια. Διότι φαίνεται πως δεν αρκεί αυτό που κάνουμε ήδη. Δεν αρκεί να δίνουμε μόνο χρήματα για την, ε, τον εξοπλισμό της βιομηχανίας τους και τα λοιπά. Χρειάζονται περισσότερα πράγματα. Είναι τόσα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει η Αφρική και τελικά φτάνουμε και σε ε, παραδείσους φορολογικούς. Όλα αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Ευχαριστώ κύριε Μάνκα. Κύριε Φιντά αν έχετε την καλοσύνη. Έχετε το λόγο Μην απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ εύτοχες ερωτήσεις στα γαλλικά. Ε, δεν τις ακολουθώ με τη σειρά που ακούστηκαν γιατί πολλές είναι κοινέ. Ξεκινώ με αυτό που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, ότι πρωταρχικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το, τη δημογραφική πρώτη πρόκληση. Ένα-δύο δισεκατομμύρια τώρα, το 2050, εάν ε, αν ευσταθούν οι προβλέψεις που κατά πάσα πιθανότητα ευσταθούν, 2,4 δις. Πίεση δηλαδή για τις κοινωνίες, τις οικονομίες αυτές, πραγματική πίεση. Και βεβαίως, εάν δεν μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε μια θετική δυναμική από την Αφρικανική Ήπειρο. Οι συνέπειες, το spillover για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι τεράστιες ανεξαρτήτως του τι θα κάνουμε για να ελέγξουμε την, την οδό της Μεσογείου. Κινητοποίηση λοιπόν, πολιτική κινητοποίηση, μίζων, χρειάζεται, απαιτείται και απαιτείται τώρα. Όπως είπατε, χρειάζεται μια γνήσια πολιτική εταιρική σχέση που να αλλάζει τα δεδομένα, να αλλάζει στάση σε σχέση με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, σας δεκόπτω. Μας είπατε τώρα ότι με τις, προκλη... με τις προβλέψεις θα έχει 2,4 δις το 2050 η Αφρική. Δηλαδή το... σε σχέση με, με τον τωρινό πληθυσμό. Ε, τα διπλάσια κύριε πρόεδρε. 1,2. Τώρα 2,4 το 50. Άρα το 2050 η Αφρική θα είναι η πολυπληθέστερη περιοχή και η περιοχή με τον πιο ηλικιο, με το πιο νεαρό πολιτισμό, ε, πληθυσμό του κόσμου. Όλες οι ήπειροι πλην της Αφρικής. Άρα χρειάζεται πολιτική στράτευση και αλλαγή στάση και νοοτροπίας ουσιαστική σε σχέση με αυτά που έχουμε υπόψη τώρα. Δηλαδή τη σχέση δωρητή και αποδέκτη της δωρεάς. Και σε αυτό ακριβώς στέκομαι, όπως είπα και νωρίτερα, ότι τα ποσά που διαθέτουμε θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με ένα πολιτικό θεματολόγιο συγκεκριμένο ή σύνοδος της Αμπιτζάν. Σε αυτό θα σταθεί και εμείς έχουμε επιμείνει από πλευρά μας αλλά και τα κρατημέλη ιδιαίτερα στην ιδέα ότι για να περπατήσει κανείς, για να πω το παραλληλισμό που βρίσκω πιο εκφραστικό, χρειάζονται δύο πόδια. Δηλαδή και εμείς πρέπει να κάνουμε προσπάθεια, αλλά την αντίστοιχη προσπάθεια πρέπει να κάνουν και οι Αφρικανοί εταίροι. Και θα το εκφράσει αυτό ο Ρομπέρτο, ε, γιατί μεταφράζεται στον οικονομικό τομέα πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή πρέπει η Αφρική να κάνει περισσότερες επενδύσεις από ό,τι τώρα και εμείς από πλευράς μας μπορούμε αξιοποιώντας την αναπτυξιακή βοήθεια να ε, εξασφαλίσουμε το de-risking, τη μείωση του επενδυτικού κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα και οι Αφρικανοί φίλοι μπορούν και εταίροι μπορούν να βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα. Δύο πόδια πρέπει και τα δύο να περπατάνε με τον ίδιο ρυθμό Ιδάλω δεν θα φέρουμε κανένα αποτέλεσμα. Αυτές είναι οι προτάσεις μας, οι προτάσεις ε, και για την αναπτυξιακή βοήθεια που θα υιοθετηθούν στην Αμπιτζάν. Τώρα όσον αφορά την απασχόληση. Με τη δημογραφική ανάπτυξη που έχει, η Αφρική θα πρέπει κάθε χρόνο να δημιουργεί 18 εκατομμύρια θέσεις εργασία. Καινούριε θέσει εργασία. Τεράστιο νούμερο, προφανώ μη εφικτό. Αλλά για να δημιουργηθούν στο δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας θα πρέπει να αναπτυχθεί μία δράση επενδυτική, να εξασφαλιστεί μια οικονομία προστιθέμενης αξίας και σε αυτό θα βοηθήσει το EIP και να καταρτιστούν οι άνθρωποι. Έχετε το δίκιο σε αυτό. Δεν αρκεί να δημιουργούμε θέσει εργασία. Πρέπει οι νέοι Αφρικανοί να σε θέση να τι αναλάβουν αυτέ τι θέσει εργασία και να εργαστούν. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση και στην εκπαίδευση και βεβαίως και πάνω απ' όλα στην επαγγελματική κατάρτιση. Δύο θεμελιώδεις άξονες που βεβαίως θα προωθήσουμε κατά την Σύνοδο. Και περνάμε βέβαια σε ένα πολύ λεπτό θέμα, λεπτό μεν πρέπει όμως εγώ να το θίξω, του οικογενειακού προγραμματισμού της ε, αναπαραγωγικής υγείας και των ε, δικαιωμάτων των αναπαραγωγικών. Θέμα λεπτό για ορισμένα κράτη-μέλη. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να μειωθεί η, η δημογραφική ανάπτυξη, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει χάρη στην ε, κατάρτιση των γυναικών και των κοριτσιών, χάρη στη δημιουργία θέσεων εργασία για τις γυναίκες, χάρη σε μέτρα οικογενειακού προγραμματισμού και έτσι μπορεί να μειωθεί η ε, καμπύλη ανάπτυξη ε, του πληθυσμού. Για όλα αυτά, και συμφωνώ μαζί σας, χρειάζεται δράση συλλογική, σαφέστερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Γνωρίζουμε ποια είναι τα όρια των δυνατοτήτων μας. Οι συζητήσεις για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν ε, οδηγούν σε αποτέλεσμα ικανοποιητικό, μειώνεται ουσιαστικά η εξωτερική δράση, ε, η συζήτηση για την ενσωμάτωση στον προϋπολογισμό του ΦΕΔ είναι κομμάτι αυτής της συζήτησης με όλες τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που εξήγησατε κι εσείς. Ταυτόχρονα όμως και η από κοινού διαχείριση των δράσεων μας, της εξωτερικής δράσης, σημαίνει ταυτόχρονα και τη συνεργασία, το συντονισμό, στα ποσά που διαθέτουμε στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, αυτό που ονομάζουμε κοινή κοινό προγραμματισμό. Πράγμα το οποίο ίσω να είναι δύσκολο γιατί είναι διαφορετική η προγραμματική κύκλη. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα, πολιτικό διακύβευμα και πρέπει στο μέγιστο δυνατό βαθμό η Σύνοδος Κορυφής του Αμπιτζάν και όλες οι δεσμές που θα αναλάβουμε τα κράτη-μέλη θα εκπροσωπούνται σε ύψιστο επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, κάποια άλλα σε επίπεδο υπουργών των εξωτερικών όταν, αναλάβουμε, όταν αναλαμβάνουμε κοινέ ε, δεσμεύσεις θα πρέπει και εμείς μετά, μετά τη Σύνοδο μαζί με τα κράτη-μέλη να κάτσουμε και να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων που δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά με τα χρήματα που έχουμε στη θέση μας από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό αλλά μέσα και από τους προϋπολογισμούς ε, από τους αναπτυξιακούς που διμερώς διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη και έτσι φτάνω στο τελευταίο σημείο και την παρατήρηση του κύριου Ντεπρέ που βέβαια είναι πολιτικού χαρακτήρα, αφορά πολιτική επιλογή. Είναι πραγματικό το ποσό που προσφέρει στην Αφρική η ομογένεια. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε καταρχάς για να μειώσουμε το κόστος των εμβασμάτων. Γιατί ήταν ναι, στο παρελθόν τεράστιο το κόστος αυτών των εμβασμάτων που έστελναν ε, οι ομογενείς ε, Αφρικανοί της χώρες τους, οικογένειές τους. Μετά πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα τι γίνεται, να δούμε αν υπάρχουν μέσα για να μπορέσουμε αυτά τα ποσά να τα καταγράφουμε τροποντινά ώστε να, να μην θεωρούνται τα ποσά αυτά εντάξει ένα χαρτζιλί και ένα συμπαθητικό ποσό πούμε, για προσδιάθεση είναι ελεύθερη αλλά εάν υπάρχει και τρόπος το χρήμα αυτό να διοχετευθεί για να ικανοποιήσει στόχου πιο αποδοτικούς, πιο ικανοποιητικού, ω προς τις επενδύσεις. Βέβαια είναι λεπτό το θέμα γιατί πρόκειται για ιδιωτικό χρήμα, ανήκει σε ιδιώτε. Αλλά μια προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή ασφαλώ χρειάζεται. Άρα, μια και, μια ήταν ισότιμα τα ποσά, 21 δι το 2015, εμβάσματα και 21,4 από την ε, δημόσια βοήθεια για την ανάπτυξη, όπως είπα το 2015, αν μπορεί να τα καταστήσει το ένα πόσο το άλλο, όχι δεν νομίζω. Γιατί είναι πολύ περιορισμένε οι δυνατότητε υποδοχή σε νόμιμη μετανάστευση καταρχά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενό αφετέρου, η χρήση στην οποία προορίζονται τα ποσά αυτά δεν είναι ίδια. Και εδώ η αναπτυξιακή βοήθεια, η δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια έχει τεράστια πλεονεκτήματα να προσφέρει σε σχέση με τα ιδιωτικά εμβάσματα σε ύψο 21 δισεκατομμυρίων. Ε, σε όρους βιώσιμης ανάπτυξης ε, ε, των χωρών αυτών της Αφρικής είναι πολύ πιο αποδοτικές, ε, πιο αποδοτικά τα 21,4 δι της δημόσιας αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά και ευχαριστώ, Ελπίζοντα ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας. Ο Πρόεδρος, ναι, απαντήστε τόσο καλά που θα διατυπώσουμε και άλλες ερωτήσεις από ό,τι φαίνεται. Διαδραστική συζήτηση, κύριε Ντεπρέ. Ναι, ήταν λίγο προκλητική η ερώτησή μου, αλλά είχε ένα συγκεκριμένο νόημα πιστεύω ότι με την τωρινή δημογραφική έκρηξη και πιστεύω ότι θα αλλάξει, θα μειωθεί το επίπεδο γεννητικότητα με την ανάπτυξη της ε, απασχόλησης και της εκπαίδευση πάνω απ' όλα, μήπως θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την πίεση στη μεταναστευτική ροή. Ίσως αυτό να τρομάξει κάποιους, αλλά Πιστεύω ότι με όλα τα μέσα που έχουμε κινητοποιήσει δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τις, δημογραφικές, τις μεταναστευτικές ροές, ιδιαίτερα από την υποσαχάρη Αφρική. Δεν το πιστεύω που δεν είναι αυτή. Και αυτό και βέβαια γιατί υπάρχει δημογραφική πίεση, αλλά και γιατί πλέον υπάρχουν και οι κλιματικές πιέσεις, οι πιέσεις της κλιματικής αλλαγής. Επίσης έχω να πω ότι αν κάποιος έχει έρθει από εδώ και πάει εκεί, το χρήμα αυτό αφορά ιδιώτη, έτσι στέλνει χρήμα, αφορά ιδιότητα, ένα χρήμα το οποίο διατίθεται ιδιωτικά χωρίς ανάγκη ε, γραφειοκρατικών ε, δομών που παρεμβαίνουν. Δηλαδή μια οικογένεια παίρνει τα χρήματα του εμβάσματος, πάει στο γιατρό κτλ. Μην το υποτιμούμε αυτό, τη σημασία του. Ήθελα να το συζητήσουμε αν υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν μηχανισμοί που να επιτρέπουν κάτι πιο συλλογικό σε κάποια στιγμή μια βοήθεια αναπτυξιακή πιο ουσιαστική και επίσης αυτή η πληθώρα μέσων που υπάρχουν και στα εθνικά κράτη και στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, μέσα ή εντός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, συνιστούν μια απίστευτη απίστευτα βαριά γραφειοκρατική δημή. Μα κάτι πρέπει να αλλάξουμε και στην οτροπία μας και στην πολιτική μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να, και να συνεχίσουμε όλοι μαζί, ελπίζω. Ο πρόεδρος. Δηλαδή, θέλετε, ένα αμφιβόλο το οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Τεπρέ. Θα έπρεπε να γίνει μια καλή ε, ελεγκτική δραστηριότητα στο οργανόγραμμα της Επιτροπής. Ο κύριος Φερνάντες και μετά, Φερνάντες, και μετά ο κύριος Κολμέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική συζήτηση. Εγώ θα δώσω την έμφαση στη σημασία της παιδείας. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις χωρίς να κάνουμε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται ε, καιρός για να γίνει κάτι τέτοιο. Η ερώτησή μου είναι, έχουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ενδιαφέρονται ήδη ε, ε, χώρες, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενες χώρες. Ε, αυτό είναι επειδή λειτουργεί με πλατφόρμες. Ε, πότε πιστεύω ότι θα αρχίσει να χρησιμοποιείτε, δηλαδή πότε θα αρχίσει να εκτελείτε Μέσα σε αυτό το πολιτές ή μετά. Και ακόμα και αν είναι στο επόμενο πάλι καλά θα είναι. Και επίσης και με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ποια είναι το χρόνο διάγραμμα εκτέλεσης. Θα είναι και το δεύτερο τμήμα σε λίγο. Ναι, ναι, αλλά απλά ε, προχωρώ λίγο την εργασία. Κύριε Σκόλμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να κάνω μια υπερώτηση. τα σύντομα πριν από έξι μήνες είχα την ευκαιρία να πάω ε, στην Αφρική και να εκπροσωπώντας ε, μια τραπέζα στην Αφρική λοιπόν η σημασία δεν είναι να δούμε μόνο τα χρήματα που μπαίνουν αλλά ε, και το να υπάρχουν σταθερά κράτη στα οποία επενδύει κανείς τα χρήματα, γιατί αλλιώς ε, ε από το ποσό για το οποίο μιλάμε, ε, πάνω στον κάδο τα χρήματα και καλό θα ήταν να μην ε, ε, γίνεται αυτό γιατί δεν βλέπουμε τις δομές που τελευταία θέλουμε και ο καθένας μπορεί να λέει ότι ε, θέλει να κάνει κάτι με αυτά τα χρήματα, όμως στην ουσία υποστηρίζουμε τις υφιστάμενες ε, δομές ε, και φυσικά θα ήταν μάλλον ουτοπικό να πιστεύουμε ότι σε μία νύχτα θα αλλάξουν όλα στην Αφρική και όλες οι δομές και οι υποδομές. Καλό θα είναι λοιπόν να ακούσουμε αυτά που είπε ας πούμε ένας καθηγητής στη Γερμανία που γνωρίζει το θέμα ότι χρειάζεται τουλάχιστον 20 χρόνια ε, δραστηριοποίησης για να μπορέσουμε μετά από 20 χρόνια να έχουμε την αλλαγή. Είναι μάλλον ουτοπικό να περιμένουμε ε, μέσα σε λίγα χρόνια να αλλάξουμε την δημογραφική εικόνα. Ε, τουλάχιστον 20 χρόνια χρειάζεται για να γίνει αυτό. Να επανέλθω σε αυτό το θέμα το δημογραφικό. Είπατε από 1,5 δις στο 2,5. Ποια είναι ε, η αντιστοιχία η μάλλον η κατανομή ανάμεσα στο Μαγκρέμπ και την ε, Ποσαχάρη Αφρική. Ναι. Ε, Τώρα, ε, πιστεύω πως υπάρχουν ναι, κονδύλια τα οποία πάνε στην Αφρική και προέρχονται από την εργασία, αλλά υπάρχουν και κονδύλια που προέρχονται από την δημόσια βοήθεια, τα επιδόματα. Έχω συγκεκριμένες περιπτώσεις υπόψη μου, όπου από τις, ε, τα επιδόματα που παίρνουν Αφρικανοί τα στέλνουν κατευθείαν στην Αφρική ή ένα μεγάλο μέρος αυτών. Ε, και Όσον αφορά αυτά τα εμβάσματα που φεύγουν από την Ευρώπη προς την Αφρική, έχετε καμιά ιδέα για το τι παίρνουν οι τράπεζες που τα μεταφέρουν, οι ενδιάμεσοι. Και μήπως ε, θα έπρεπε ε, να γίνουν δημόσια αυτά, αυτές οι δίωδοι εμβάσματων, ώστε να μην υπάρχουν πλέον προμήθειες εκεί. Ναι, Πρόεδρε, ε, φεύγει πάρα πολύ χρήμα από την Αφρική όμως ταυτόχρονα παράνομα, παράνομες ροές, χρηματοοικονομικές που ξεπερνούν τα ποσά που στέλνουμε εμείς και επενδύουμε για την αναπτυξιακή βοήθεια έως και 50 δις δολάρια έφυγαν παράνομα από την Αφρικανική Ήπειρο το 2016. Και δυστυχώς συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό οι πολυεθνικές με έδρα το, την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Γκλένκο παραδείγματι η οποία για το τσάτ συγκεκριμένα έδειξε ε, ψευδή στοιχεία ως προς τα κέρδη, ποσά που φύγανε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καλύψει αναπτυξιακή βοήθεια. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε, κύριε Διευθυντά. Ναι, το λόγο τον έχω, τις απαντήσεις δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τη συμβουλή της Παγκόσμιας Τράπεζας την οποία συμμεριζόμαστε ότι δεν φτάνει η ποσότητα πρέπει να δουλέψουμε και για την ποιότητα των κρατών των εταίρων μας. Είναι εξαιρετικά παρόν στην δική μας προσέγγιση. Ο Ρομπέρτο σίγουρα θα το αναπτύξει περισσότερο γιατί θα μιλήσει για τις επενδύσεις. Εγώ αναφέρθηκα όμως στη διαδικασία εφαρμογή που θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη και είναι η δημοσιονομική στήριξη. Ποιο είναι το μεγάλο πλονέκτημα της ε, δημοσιονομικής στήριξης. Η δημοσιονομική στήριξη συνοδεύεται ακριβώς από έναν διάλογο πολιτικό θεμελιώδη συνοδεύεται από μέτρα που ενισχύουν τις δυνατότητες και τις τακτικές των εταίρων μας και εδώ αναφέρομαι και στο σχόλιο του κ. Τζέλλαρ ότι συχνά δηλαδή εκεί περιλαμβάνονται σημαντικά στοιχεία δημόσια, ε, διαχείρισης δημόσιας ε, ε, οικονομίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η νέα ατζέντα θα αναφέρεται ιδιαίτερα στη κινητοποίηση των εγχώριων πόρων. Domestic Resource Mobilization. Σημαίνει αυτό απαραίτητα ε, συστήματα δημόσιας χρηματοδότησης που είναι πολύ σταθερά. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε επιθετική ε, ατζέντα για να καταπολεμήσουμε τις παράνομες ε, δημοσιονομικές, ε, χρηματικές μάλλον ροές. Το είναι πρόβλημα για την Αφρική, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε μια διαρροή κονδυλίων που πρέπει οπωσδήποτε να πάψει. et ça devient en plus une priorité ε, και αυτό γιατί σημαίνει ότι και αυτό το θέμα μάλλον έχει έρθει στο επίκεντρο του διεθνούς θεματολογίου της Ατζέντα 2030 δηλαδή. Από αυτή την άποψη λοιπόν συμφωνώ απόλυτα ότι η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε σε σχέση με την Αφρικανική Ήπειρο είναι μακρόπνοη. Οι μεταναστευτικές πιέσεις ή το δημογραφικό διακύβευμα δεν είναι κάτι που ρυθμίζεται εντός 2-3 ετών, ούτε καν εντός πενταετίας. Πέρα από εκεί θα πρέπει να δεσμευτούμε για πιο μακροπρόθεσμα Ξού και η σημασία των όσων έχουμε φτιάξει για το καταπίστευμα το μεταναστευτικό για την Αφρική. Ε, στόχος είναι να διευκολυθούν οι έρευνες που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε καλύτερα τι είδους παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε με κάποιο αντίκτυπο, ελπίζουμε, και έχουμε φτιάξει ανεξάρτητα ένα σύστημα παρακολούθησης που στη συνέχεια θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε αν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε έχουν το αναμενόμενα αποτελέσματα, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί τα, η δουλειά πάνω στις βαθύτερες αιτίε της μετανάστευσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας καθοδηγήσει για το μέλλον. Άρα λοιπόν πρέπει να, στο πλαίσιο του προγραμματισμού για τον επόμενο κύκλο, το επόμενο PDP, θα πρέπει αυτά όλα να τα λάβουμε υπόψη με περισσότερες λεπτομέρειες. Επί τη βάση αυτής της ερευνητικής δουλειάς που έχουμε ξεκινήσει. Για το θέμα της Αφρικανικής Διασποράς δεν έχω νούμερα. Δεν μπορώ να σας δώσω νούμερα ακριβώς για το ποια είναι η σύσταση της προέλευσης αυτών των ευασμάτων, σε ποιο βαθμό δηλαδή είναι χρήματα που έχουν, έχει κερδίσει η διασπορά μέσω της εργασίας της ή αν είναι από τα επιδόματα που παίρνουν ορισμένοι μετανάστες που διαμένουν νομίμω στην Ευρώπη και μετά τα μεταβιβάζουν. Εν περιπτώσει αυτό τις λεπτομέρειες δεν τις έχουμε. Ε, διερωτόμαστε, μπορούμε να ρωτήσουμε μήπως και τα καταφέρουμε να έχουμε αυτή τη δεν πρέπει να είναι και τόσο προφανές, αλλά πάντως ένα τμήμα της δημόσιας αναπτυξικής βοήθειας που εμείς συμμετράμε δαπανάται και στην Ευρώπη που χρησιμοποιείται για την υποδοχή ακριβώς των προσφύγων στην Ευρώπη. Ένα τμήμα της αναπτυξιακής βοήθειας λοιπόν Ποιο κομμάτι ρωτάει ο πρόεδρος. Γιατί κάποιες φορές δεν το καταλαβαίνουμε καλά πόσα χρήματα. Λέτε λοιπόν ότι από τα 21,5 δις ένα κομμάτι χρησιμοποιείται για την υποδοχή των προσφύγων εδώ. Μάλιστα, είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, όταν βλέπουμε νούμερα, αλλά όταν πάμε να τα δούμε από κοντά υπάρχει ανακύκλωση και Καλοπισμός. Όχι καλοπισμός, γιατί είναι δηλωμένα όλα αυτά ετησίως, πολύ ξεκάθαρα στον ΩΣΑ, στο, που κρατάει πολύ ξεκάθαρα στοιχεία ε, και για τα διάφορα κριτήρια τα οποία μπορούμε να λάβουμε υπόψη. Στον που είναι DAC, Μπολόλα, είναι στο ντάκ. Ε, Αυτά σίγουρα θα σας τα δώσουμε, βεβαίως, τα έχουμε. Και αυτό με, φτάνει, με φέρνει στο σημείο, στην παρατήρηση του κ. Ντεπρέ, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ευάσματα. Να συμπληρώσω. Πρόκειται όντως για ποσά ατομικά μεμονωμένα, τα οποία συχνά ε, ε, εμβάζονται στις οικογένειες αλλά όλα είναι και περισσότερο βλέπουμε ότι αυτά τα ποσά χρησιμοποιούνται για επενδύσεις που δεν αφορούν μόνο μία οικογένεια, αλλά χωριά, κοινότητες. Το βλέπουμε ας πούμε στην Σομαλία. Εντάξει, τώρα περνά πιο δύσκολη κατάσταση η χώρα, αλλά βλέπουμε ότι η Σομαλία προσπαθεί να ξαναγεννηθεί ως κράτος και όπου η διασπορά που είναι πολύ σημαντική στην Ευρώπη, στον Καναδά και στη ΗΠΑ, αρχίζει να κινητοποιείται. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για έμβασμα χρημάτων στην οικογένεια που βρίσκεται ακόμα εκεί, αλλά για μια πραγματική πολιτική ε, που έχει επιρροή στην ανάπτυξη κάποιων χωριών, πόλεων, λιμανιών. Βλέπουμε λοιπόν χρήσιμη χρήση αυτών των ε, χρημάτων. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Φερνάντες ότι είναι ουσιώδους, ε, ουσιώδες ε, και θα πρέπει να επανέλθουμε δυναμικά στον τομέα της παιδείας και της κατάρτισης. ήδη έχει μεγάλη σημασία, αλλά θα ε, πάρει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην αναπτυξιακή βοήθεια μετά το 2020. Για τη Γαλλία, το έχουμε σαφώς, ε, η Γαλλία το έχει σαφώς αναφέρει όσον αφορά την Αφρική. Να πω ε, τώρα, άλλη μια φορά θα σας απογοητεύσω κύριε Πρόεδρε για τα στοιχεία της διαφάνειας, της τα δημογραφικά και την κατανομή ανάμεσα στη Βόρεια Αφρική και την Υποσαχάρη Αφρική δεν ξέρω τα στοιχεία απ' έξω, πάντως μπορώ να σας τα στείλω και να, σας τα... να τα βρω και να σας τα στείλω αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στο προπολογισμό 2018 που μόλις ολοκληρώθηκε με τη συνδιαλλαγή του Σαββάτου προβλέπεται ένα ποσό με πρόγραμμα έρασμους για νέους που έχουν δεξιότητες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αγρονομικές να παρακολουθήσουν την εκτέλεση των κονδυλίων που είναι αφιερωμένα στο πλαίσιο της ε, βιώσιμης, ε, της ε, βιώσιμης ανάπτυξης για την Αφρική. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρομπέρτο Ριντόλφη πρέπει να πω ότι έχει το πολύ σημαντικό τίτλο «Διευθυντής του πλανήτη και της ευημερία. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Είναι ένας, πραγματικά, ένας τίτλος ο οποίος πραγματικά με υποχρεώνει σε μεγάλα έργα. Ε, σας ευχαριστώ καταρχάς για την υποδοχή σας εδώ. Ευχαριστώ εσάς προσωπικά κύριε Πρόεδρε για την βοήθεια που προσφέρατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της ε, επεξεργασίας του μέρους διαλόγου για το Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όλα αυτά που είπατε τώρα πρέπει να μετατραπούν σε πραγματικότητα. Γι' αυτό πριν από 1,5 χρόνο περίπου επεξεργαστήκαμε την ιδέα ενός εξωτερικού προγράμματος επενδύσεων κάπως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που υιοθέτησαν το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο. Το Ταμείο είναι το κομμάτι που διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, το είπατε και εσείς, και γι' αυτό υπάρχουν τρεις πυλώνες. Πριν όμως προχωρήσω στην ε, παρουσίασή μου που θα έρθει στα αγγλικά, επιτρέψτε να πω ένα-δυο λόγια εισαγωγικά. Πρέπει να προχωρήσουμε πάνω στη γραμμή των ε, policy decisions, των αποφάσεων ε, πολιτικών επιλογών και όχι σε επενδύσεις. Το είπαμε και πριν, εμείς προσπαθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενώσουμε τα ταμεία γιατί οι πολιτικές επιλογές, ε, το έργο που έχουμε να έχει έχουν πρωταρχική σημασία και μετά βεβαίως έχουμε γραφειοκρατικές δομές στα ταμεία δυστυχώς, αλλά αλλά εγώ σας εκλυπαρώ. Στο μέλλον ό,τι δομές παρακαλώ να είναι πιο απλές. Δεύτερον, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις. Θα θυμάστε ασφαλώς μια ανακοίνωση του 2014 που είχα συντάξει, γιατί εγώ είμαι ο ειδικό της υβριδοποίησης ε, της αναπτυξιακής βοήθειας, η ειδικότητά μου η υβριδοποίηση. Και είχαμε μια πολύ καλή ανταπόκριση το 2014 από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προς το ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό αποτελεί μια πολιτική βάση για να προχωρήσουμε μετά πιέζοντας ιδιαίτερα με συγκεκριμένα μέσα. Ε, η Αφρικανική Ήπειρος και συμφωνούμε όλοι, η δημιουργία θέσεων εργασίας για την Αφρικανική Ήπειρο είναι πρωταρχική προτεραιότητα για όλους αυτούς τους λόγους που εκθέσατε εσείς. Αλλά τις θέσεις εργασία. Ποιο θα τις δημιουργήσει. Όχι πάντως οι κυβερνήσεις. Οι επιχειρήσει, ναι. Και άρα τίθεται εδώ το πρωταρχικό ερώτημα. Υφίσταται περιβάλλον για την αναπτυξιακή βοήθεια. Και δύο λόγια ακόμη για τους ομογενείς, για να συνεχίσουμε μετά με την συζήτηση και την παρουσίαση, μετά τη σύντομη αυτή εισαγωγή. Η ομογένεια, ναι, αλλά, αλλά πρόσοχη, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα μια συνιστόσα την οποία δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε. Είπε ο συνάδελφο ότι έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια για να μειωθεί το κόστο των εμβασμάτων. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε ότι είχαμε τη Western Union και όλα αυτά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ήταν τεράστια τα τέλη ε, για το έμβασμα. Όσο πιο μικρό ήταν το ποσό του εμβάσματο, τόσο μεγαλύτερη και η χρέωση. Ανήθικο, ανήθικα επίπεδα χρέωση. Έχουμε μειώσει σημαντικά, όχι όμω τα επίπεδα που θα θέλαμε. Αλλά όταν έχουμε να κάνουμε από, για εμβάσματα από ιδιώτη σε ιδιώτη. Δεν το καν να το συζητούμε, όχι να το ακουμπήσουμε, γιατί είναι κάτι που εγώ θα δώσω στην οικογένειά μου. Για τις ανάγκες της, για όποιες ανάγκες της. Από την άλλη, ο μετανάστης στην Ευρώπη παράγει πλούτο και αυτό το πλούτο καμιά φορά τον επενδύει και στα ομόλογα του κρατικού ταμιευτηρίου, της, ε, ταχυδρομικού ταμιευτηρίου της Γερμανίας, της Γαλλίας, κάπου Πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη λοιπόν. Γιατί πολλές φορές και τα συνταξιωτικά ταμεία, ο ιδιώτης επενδύτης, έχει την ευκολία να αναλάβει ένα κίνδυνο χωρίς να κινδυνεύει το κεφαλαίο του. Να κάνει μια επένδυση χωρίς να κινδυνεύει το κεφαλαίο του. Για να δω αν μπορώ να βάλω μπρος αυτές τις διαφάνειες. Ωραία. Πού να το πουντάρω αυτό το, φέκι, λέει ο Πούντε. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν τα SDGs είναι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ε, και είμαστε πιστοί σε αυτούς τους στόχους ε, γιατί δεν είναι μόνο θέμα αύξησης του ΑΕΠ αλλά και του περιβάλλοντος ε, και της ταχύτητας των επενδύσεων. Θα γυρίσω τώρα στα αγγλικά. Euh, Έχουμε ένα ε, παγκόσμιο πλαίσιο ε, μέσα στο οποίο ορίζεται αυτό το σχέδιο. Είναι η ατζέντα δράσης της Αντίς Μπέμπα. Τον Ιούλιο του 2015 αποφασίστηκε ότι ε, το όντι από μόνο του δεν είναι αρκετό, γι' αυτό κάνουμε μόχλευση των χρημάτων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη εγκρίθηκε και εδώ έρχεται και ο τίτλος μου, τα 5 P. People, Peace, Prosperity, Planet and Partnership. Οι άνθρωποι, η ειρήνη, η ευημερία, ο πλανήτης και η εταιρική σχέση. Αυτή είναι η στρατηγική μας, η παγκόσμια στρατηγική και η πολιτική ε, ο πολιτικός προσανατολισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον εξωτερικό κόσμο. Ε, προσπαθούμε να είμαστε εκεί και να τους περιλαμβάνουμε όλους. Θα θυμάστε κύριε Πρόεδρο πριν από 50 χρόνια δεν μας επιτρεπόταν καν να συζητούμε τα συμφέροντά μας. Η αναπτυξιακή πολιτική ήταν μια μορφή ε, Πάμε τώρα στην, ε, στους στόχους ε, της βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη, στις δουλειές, ε, στις θέση εργασίας δηλαδή, το περιβάλλον, την ε, διαφθορά που δεν είναι εύκολο. Ήμουν πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας από τους παράγοντες ε, που δεν ενθάρρυναν τους επενδυτές ήταν αυτή η γραφειοκρατία και η διαφθορά. Όσο περισσότερες είναι αυτές, τόσο ε, πιο δύσκολες οι επενδύσεις, γιατί πρέπει να ασχολείσαι και με περισσότερο χώρο, κόσμο. Και όλα αυτά είναι πράγματα που ε, δυσχεραίνουν την διαδικασία. Πριν από 1,5 χρόνο, όταν ε, συντάχθηκε αυτό το έγγραφο, δεν υπήρχε διέξοδος και μάλιστα τα χρήματα ακόμα και σήμερα είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις ανάγκες. Χρειαζόμαστε 210 δις το χρόνο περισσότερες επενδύσεις κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να πάμε προς τους ε, στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης που είναι ε, να συμπεριλαμβάνονται όλοι, να είμαστε βιώσιμοι και φιλικοί στο περιβάλλον το σχέδιό μας ε, για την εξωτερική δράση δεν καλύπτει όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εξωκόσμο, δηλαδή τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, την Κεντρική Ασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την Αφρική και την γειτονία. Τώρα, οι τρεις πυλώνες. Πρώτος πυλώνας, το Ταμείο. Να σας πω ότι με την η υπογραφή του Προέδρου το, στις 27 Σεπτεμβρίου θέσαμε σε ισχύ το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στις 28 έγινε η πρώτη συνάντηση με τους εισηγητές, με τον επικεφαλής ε, της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης ε, για τους στρατηγικούς στόχους του Ταμείου. Στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 7 Νοεμβρίου είχαμε την πρώτη συνάντηση του Επιχειρησιακού Συμβουλίου με τα παράθυρα που θα δείξω. Άρα, έχει δημιουργηθεί αυτό το ταμείο, το οποίο έχει δύο κομμάτια, το παραδοσιακό blending. Δίνουμε επιδοτήσεις για να μπορέσουμε να μειώσουμε το βάρος των ε, δανείων για τις δημόσιες επενδύσεις όπως είναι τα έργα τα οδικά, οι γραμμές μεταφοράς ενέργειας, ε, φωτισμός το blending το κάνουμε εδώ και 10 χρόνια. Από το 2007 έως το 2016 στην Αφρική χρησιμοποιήσαμε γύρω στα 2 εκατομμύρια ε, επιδοτήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε ε, στον δημόσιο τομέα περισσότερες υποδομές, δημόσιες επενδύσεις. Στην περίοδο 2007-2016 ε, δεσμεύσαμε 1,2 δις και από αυτά είχαμε επενδύσεις ύψους 13 δις, δηλαδή ε, το κλάσμα είναι 1 προς 11. Λειτουργεί λοιπόν αυτή η μη επιστρεπτέα ενίσχυση που δίνουμε. Είναι 10 χρόνια blending και ανάπτυξης που έρχεται ε, μέσα από τα δάνεια, από τράπεζες όπως η ΕΤΕΠ, η Αφρικανική ε, Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και από άλλους διμερείς ε, εταίρους, από τη Γαλλία κτλ. Όλα αυτά δίνουν μια όθηση σε αυτή την επιχειρησιακή δράση τώρα. Για την ε, χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα έχουμε την εμπειρία, έχουμε τα δεδομένα. Στο ελεγκτικό συνέδριο μάλιστα υπερασπίστηκα την Κομισιόν όταν μας έκαναν έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο για το blending πριν από 1,5 χρόνο και ήταν όλα πολύ θετικά. Φυσικά υπήρξαν συστάσεις για βελτίωση, αλλά το κομμάτι της ε, εγγύησης για τις ιδιωτικές επενδύσεις για τη μείωση του ρίσκου ήταν κάτι καινούριο. Γι' αυτό έπρεπε να εγκρίνουμε τον ε, κανονισμό, ο οποίος για πρώτη φορά δίνει αυτή την ε, ευθύνη για τα έκτακτα στο μεγάλο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα ποσό 700 εκατομμυρίων, 750 εκατομμυρίων. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας, η προετοιμασία των επενδύσεων από τους ιδιωτικούς ε, φορείς και τους δημόσιους φορείς και υπάρχει και ο τρίτος πυλώνας που είναι το επενδυτικό κλίμα, οι μεταρρυθμίσεις, η πατάξη της διαφθοράς, η διασφάλιση ότι κάθε χώρα έχει την δυνατότητα να δίνει την να περισχύει το κράτος δικαίου μέσα από τις κατάλληλες δικαστικές δομές και διαδικασίες. Επίσης, έχουμε μια μεγάλη καινομονία να σας πω ότι οι συνάδελφοι στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσιγκτον εντυπωσιάστηκαν και ήμασταν περήφανοι και εσείς να είστε περήφανοι γιατί για πρώτη φορά εδώ ε, ήμασταν καινοτόμοι και στην Ουάσιγκτον ε, εξεπλάγησαν γιατί αυτή ήταν η αβανγκάρντ ε, της χρηματοοικονομικής μηχανικής και τώρα εμείς τους φτάσαμε. Ανοίξαμε και ένα παράθυρο για τον ιδιωτικό τομέα στην ΕΤΕΠ. Τώρα τι είναι η τρίτη αυτή λάμπα. Είναι οι λάμπες χαμηλών εκπομπών. Η, η τρίτη είναι το One Stop Shop. Είναι ένα web portal, ένα μικρό back office που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στην Κομισιόν για να έχουμε φιλική διεπαφή με τους ε, ιδιώτες και τις, τις επιχειρήσεις δηλαδή. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση στην Κομισιόν γιατί θέλουμε να έχουμε έναν μηχανισμό αποδέσμευσης ο οποίος ε, θα έχει να κάνει με προτάσεις από τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες ε, θα μεταδίδονται, θα δίνονται στο επιχειρησιακό κομμάτι των επενδυτικών ε, βραχιώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγγύηση ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Διάσημη Ανάπτυξη είναι ένας μηχανισμός μείωσης των κινδύνων για τη δημιουργία επενδύσεων στην Αφρική και τη γειτονία. Δεν θέλουμε να δίνουμε επιδοτήσεις εκεί που γίνονται οι επενδύσεις, θέλουμε όμως ε, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις εκεί που δεν πάνε σήμερα. Και γι' αυτό πρέπει να ε, κάνουμε το λεγόμενο credit enhancement των επενδύσεων. Ο πυλώνας 1 στις εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα δείτε και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, άρθρο 8, προσθετικότητα, δηλαδή πάμε εκεί που δεν πάει κανείς και για να το κάνουμε πρέπει να πάμε και εκεί που πάνε όλοι. Για να έχουμε την προσέγγιση τύπου φάκελος, πορτφόλιο. Δεν πρέπει να πας ε, στην κεντροαφρικανική δημοκρατία για να επενδύσεις στον ε, ιδιωτικό τομέα, αλλά στην Κένια, την Κάνα, την ε, ακτή του Ελεφαντοστού και όλα αυτά να τα κάνεις σε συνδυασμό με τα μέρη που είναι δημοφιλή γιατί θέλεις να εγγυηθεί τα κονδύλια, αλλιώς θα τα χάσεις σε πέντε μήνες. Άρα συμπληρωματικότητα με άλλες πρωτοβουλίες, ευθυγράμμιση των συμφερόντων, δίνοντας τον κατάλληλο επιμερισμό κινδύνων, οικονομική και χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα. Ε, υπάρχουν τα οικονομικά κομμάτια, αλλά υπάρχει και το κομμάτι που θέτει Κομισιόν, το, κοινωνικό, το, η επαγγελματική κατάρτιση έχουν να κάνουν με τον πυλώνα 3. Όλα αυτά εξηγούν την προσθετικότητα και όσο μπορούμε επικεντρωνόμαστε στους νέους και στις γυναίκες είναι τα προτινόμενα παράθυρα επενδύσεων που έχουν εγκριθεί, έχουν πάει στο Επιχειρησιακό Συμβούλιο και τώρα θα πρέπει να ε, εγκριθούν και από εκεί. Νομίζω αύριο θα λάβει την απόφαση η Κομισιόν. Είναι πέντε. Βιώσιμη ενέργεια και συνδεσιμότητα, μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες και μεγα... επιχειρήσεις. Εχθές μιλήσαμε για την συμπερίληψη στα χρηματοπιστωτικά. Μιλήσαμε για το microfinance. Τρία, βιώσιμη γεωργία. Εκεί περιμένουμε το μέγιστο αριθμό θέσεων εργασίας. Τέσσερα, βιώσιμες πόλεις. Πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει μεγάλη μετανάστευση από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές, χωρίς όμως επένδυση στις χώρες, στις πόλεις θα έχουμε καταστροφή. Οι πόλεις διωγγώνονται δραματικά γρήγορα και δεν υπάρχει αντίστοιχη, αντίστοιχος προγραμματισμός. Και τέλος ε, είναι η ψηφιακή ανάπτυξη. Για την ψηφιακή ανάπτυξη να πω ότι οι αγορές λειτουργούν. Υπάρχει χρηματοδότηση για τέτοιες επενδύσεις, όμως σε κάποια θέματα είναι πιο λίγες οι επενδύσεις. Γι' αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε. Τώρα, σε αυτό ήθελα να επικεντρωθούμε, στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον πυλώνα 2, την παροχή τεχνικής αρρωγής, για να μπορέσουμε από τη μία ο πυλώνας Έλλας ένα, η επένδυση πρώτα αυτοποίηση το ο πυλώνας 2, η ανάλυση της αλυσίδας αξίας και της αγοραστικής αξίας να έχουν αποτέλεσμα. Θα δούμε τώρα αυτό που θέλουμε να έχουμε σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε την ολοκλήρωση αυτών των διαφόρων τομέων. Τι ήθελα να σας εξηγήσω εδώ. Ίσως ε, καλό θα ήταν να μάθετε πώς λειτουργούν τα κονδύλια. Δεν έχω διαφάνεια, αλλά θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω με έτσι παραστατικό τρόπο. Η εγγύηση θα είναι σαν τα θεμέλια του κτηρίου θα φέρει το περισσότερο βάρος ε, του κτηρίου και το περισσότερο ρίσκο. Στο ισόγειο θα έχουμε την ε, αναπτυξιακή τράπεζα που θα βάζει τα χρήματα. Θα φέρει και αυτή ε, κάποιο ρίσκο και κάποιο βάρος, αλλά όχι όσο τα θεμέλια. Και πάνω στο... θα έχουμε 4, 5, 6, 7 ορόφους που θα είναι οι θεσμικοί επενδυτές, π.χ. συνταξιδοτικά ταμεία. Φανταστείτε 100 εκατομμύρια εγγύηση που δίνει το Ταμείο, 200-300 ε, ε, εκατομμύρια από την ε, Τράπεζα, την Αναπτυξιακή και 1,5 δις από διάφορους άλλους επενδυτές που είναι προσανατολισμένοι πιο πολύ στην αγορά, όπως τα συνταξιδοτικά ταμεία. Και εκεί μπορούν να τοποθετηθούν και κάποια από τα εμβάσματα των μεταναστών. Όχι ακριβώς τα εμβάσματα, αλλά τα χρήματα που αποταμιεύουν οι μετανάστες σήμερα μπορούν να συνδεθούν με παραγωγικό τρόπο με αυτό. Άρα η μόχλευση είναι το πρώτο κριτήριο, η προσθετικότητα το δεύτερο κριτήριο και οι δουλειές που δημιουργούνται αναμονάδα επένδυσης χρημάτων φορολογουμένων είναι το τρίτο κριτήριο. Αυτά τα τρία είναι τα πιο σημαντικά. Υπάρχουν και άλλα. Κύριε Πρόεδρε, θα σταματήσω εδώ για να δώσω λίγο χώρο για συζήτηση και ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για αυτή την πληρέστατη εισήγηση. Καταλάβαμε πολύ καλά τι θα προσφέρει το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Θα δώσω το λόγο τώρα στον Πρόεδρο Βάταρα για να μας δώσει τη δική του εκτίμηση ε, για τις ανάγκες και τους προσανατολισμούς που ακολουθούμε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτή τη τόσο ενδιαφέρουσα συνεδρίαση ε, για τους, ε, τις, για την Αφρική. Να σας δώσω κάποια στοιχεία πριν να περάσω στο οικονομικό θέμα για την προοπτική της ε, αναπτυξιακής βοήθεια. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω καταρχά όσον αφορά τη συμβολή της ε, ομογένειας. Επειδή εγώ ίδιος είμαι μετανάστης ε, πανεπιστημιακός, ε, μπορώ να εκτιμήσω τι γίνεται με την ομογένεια. Ένα μεγάλο κομμάτι της ομογένειας στην Ευρώπη επιθυμεί να επιστρέψει για να συμβάλλει στην ανάπτυξη των εκάστοτε χωρών. Αλλά υπάρχουν διάφορα εμπόδια που συναντάμε. Ένα από αυτά είναι η διακυβέρνηση. Και να σας το δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Στην, ε, ε, μέσα στο πλαίσιο των ε, ε, δραστηριοτήτων μας ε, για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση είχαμε έναν επενδυτή για, που ήθελε να επενδύσει για την κατασκευή μιας ηλιακής, ε, ενός κεντρικού μάλλον σταθμού ενέργειας, ηλιακής ενέργειας. Και αυτό το είδαμε το project, οι μελέτες μοιραστήκαμε με τους επενδυτές και μετά υπήρχαν ζητήματα πολύ πιο τεχνικά και πιο εις προσεγγίσαμε λοιπόν τις κυβερνήσεις στη Δυτική Αφρική, τα Υπουργεία, Υπουργεία Ενέργειας των ε, χωρών αυτών. Δεν λάβαμε καμιά απάντηση. Παίρνουμε απαντήσεις μετά από δύο, τρεις, έξι μήνες. Κατανοείται λοιπόν ότι ένας επενδυτής δεν μπορεί να περιμένει ε, τέτοιο διάστημα για να επενδύσει και τον κάνει να αμφισβητεί τις δυνατότητες ε, διαχείρισης της επένδυσης ε, από πλευράς ε, των όσων πάρουν αυτή την επένδυση. Με κάποια στιγμή είχα τη δυνατότητα να κάνω, έχω μια ανταλλαγή απόψεων με έναν από τους ηγέτες ε, των χωρών της Δικής Αφρικής και το είπα ότι τις περισσότερες φορές είναι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί που διαχειρίζονται τις επενδύσεις. Δηλαδή είτε γίνει επένδυση ή όχι, αυτό δεν έχει καμία, κανένα αντίκτυπο στον άνθρωπο που αναλαμβάνει το φάκελο. Κάναμε λοιπόν την εξή πρόταση. Γιατί να μην σκεφτούμε μια μεταβλητή αμοιβή αυτών των ανθρώπων που διαχειρίζονται τις επενδύσεις. Γιατί στον τομέα της πρόσβασης στις επενδύσει, Ειδικά στην Αφρική υπάρχουν ένα σωρό μεσίτε, εταιρείε, σύμβουλοι και διάβολοι οι οποίοι ε, αυτοί ε, αμείβονται για τα αποτελέσματα. Η απάντηση που λάβαμε μας εξέπληξε και κλείσαμε την πόρτα κατευθείαν είπε ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε τέτοια πρόταση. Και λίγο χρόνο μετά ο ίδιος αρχηγός κράτους μιλάει με Ευρωπαίους πολιτικούς ζητώντας περισσότερες επενδύσεις στη χώρα του. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα συνοχής, συνέπεια στην προσέγγιση. Οι άνθρωποι ομογενείς που ξέρουν καλά την, την τοπική νοοτροπία αλλά και τις προσδοκίες των επενδυτών δεν εισακούγονται από τους Αφρικανούς ηγέτες. Αυτό λοιπόν για να καταλάβουμε λίγο επίσης για την ομογένεια τα χρήματα δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που ε, επηρεάζει την μετανάστευση. Εγώ, εγώ είμαι ξένος, έχω μεγαλώσει στην Αφρική και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και η ευθύνη της επικοινωνίας. Δηλαδή τι παρουσιάζουν τα μέσα στην Αφρική, ειδικά στους νέους. μια ολόκληρη σειρά από μηνύματα τα οποία στέλνονται και επιτρέπονται από τις τοπικές αρχές και υποδηγούν τους νέους να πάρουν μια πορεία που δεν είναι καθόλου πραγματική. Δηλαδή θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε, να, να εκπαιδεύσουμε ακόμα και από το Δημοτικό και από το Λύκειο τα παιδιά να καταλάβουν, να, να, να εκπαιδευτούν στην επιχειρηματικότητα και όχι απαραίτητο να, τα όνειρά τους να είναι να φύγουν στην Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτά είναι κάποια στοιχεία λοιπόν που ήθελα να δώσω στη συζήτηση σε σχέση με την μετανάστευση. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα στοιχεία τα οποία ε, θα μπορούσαν να τονιστούν. Τώρα, για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να επανέλθω σε αυτό. Τα μέσα. Τα μέσα είναι πάρα πολύ χρήσιμα όσον αφορά την κινητοποίηση κονδυλίων. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο στο οποίο αντιμετωπίζουμε τακτικά ε, στον ιδιωτικό αφρικανικό τομέα όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Δηλαδή, το πρόβλημά μας είναι η πρόσβαση στην ενημέρωση. Τι υπάρχει ως εργαλείο, ως πίστοση, ως γραμμή επίστοσης, ως εγγύηση. Επανειλημμένα προκύπτει αυτό το πρόβλημα. Γιατί άλλο που έχουμε διαπιστώσει είναι οι πολύ περιορισμένες δυνατότητες ε, στα πλαίσια των ε, διάμεσων ε, ε, φορέων, δηλαδή τοπικές τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μια τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες και προσφέρει υπηρεσίες με βάση ένα προφίλ κινδύνου. Το προφίλ κινδύνου των μικρών και μεσαίων εταιριών δεν βρίσκει αντίστοιχε υπηρεσίε σε επίπεδο τραπεζών. Έχουμε ανθρώπου που κάποιε φορέ εγκαλούνται από τι τροπικέ τράπεζε για να αναλύσουν τα, ε, τους φακέλους. Έχουν δυσκολία στελέχωσης, δεν έχουν αρκετούς για να παρακολουθήσουν τις εταιρείε. περιορίζονται στα αιτήματα πίστοσης ε, για τις εταιρείε που έχουν πολύ καλό προφίλ κινδύνου. Έχουμε ένα παράδειγμα στην Μπουρκίνα Φάσο με ε, ένα θεσμό που δίνει εγγύησεις και έχουν λιγότερες αποτυχίες στις χρηματοδοτήσεις τους και το μυστικό είναι ότι για κάθε project που χρηματοδοτούν πάνε επί τόπου, παρακολουθούν τον διευθυντή και προβλέπουν ενδεχόμενα προβλήματα αποπληρωμής. Αυτό σημαίνει ενίσχυση των δυνατοτήτων αυτών των ε, οικονομικών φορέων. Άλλο στοιχείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θέτει στη διάθεση ορισμένων εμπορικών τραπεζών κάποιες πιστώσεις για τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα πρέπει ο καθένας να πάει σε τράπεζα. Δεν ξέρουν καν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αυτή που δίνει τα χρήματα. Δεύτερον, υπόκειται σε μια κατάσταση λες και αυτές οι τράπεζες δεν έχουν λάβει τίποτα. Πώς λοιπόν αυτοί οι ενδιάμεση τις διαχειρίζονται, διαχειρίζονται τα χρήματα, είναι στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, βραχυπρόθεσμα δάνεια, γιατί λένε ότι δεν έχουμε μακροπρόθεσμα πόρους για να παρακολουθούμε project. Μετά το κόστος των πόρων είναι στοιχεία που οι τράπεζες μας λένε έτσι, με, αυτά, με αυτές που έχουμε επαφή. Δηλαδή, και εδώ και πάλι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτή η πρόσβαση, αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα, θα πάνε σε αυτούς που τα χρειάζονται. Το καταπίστευμα τώρα να αναφέρω εδώ είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρότυπο, ώστε ακριβώς να περιοριστούν αυτές οι διαδικασίες πρόσβασης. Και ένα τελευταίο στοιχείο πριν σταματήσω θα ήταν η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Πριν από ένα-δύο χρόνια είχαμε ένα project σε επίπεδο της ομογένειας για να εντοπίσουμε τις δυνατότητες συμμετοχής της ομογένειας στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Και κάναμε ένα ερώτημα για ένα ταμείο το οποίο διαχειριζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η, Ευρω... Αφρικανική Ένωση από κοινού. Πρέπει να σας πω ότι η πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το project είχε εγκριθεί, είχε... ήταν καλό αλλά δεν μπορούσαν να απελευθερώσουν τα χρήματα από τη στιγμή που η αφρικανική πλευρά δεν είχε δώσει τη θέση της. Ε, μέχρι σήμερα δεν την έχει δώσει τη θέση της η αφρικανική πλευρά. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και τίμοι στην προσέγγιση των πραγμάτων. Το γεγονό ότι συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς είναι καλό, ναι, γιατί αναλαμβάνουν ευθύνη και υπάρχει μια αναπτυξιακή πτυχή που λαμβάνεται υπόψη, αλλά κάποιες φορές αυτό σημαίνει επιπλοκή. Ίσως θα έπρεπε να δίνεται άμεσα η πρόσβαση στους ίδιους τους επενδυτές, χωρίς την εμπλοκή των τοπικών φορέων. Des actions locales, des actions de terrain, je pense qu'ils peuvent aussi éclairer. Νομίζω πως ε, Αυτά είναι στοιχεία που επηρεάζουν την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ζητήσω στον... από την συγκέντρια. να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. <laughs> Τι βλέπει από τις πρώτες αυτές τις του Steering Board. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και τα ακούσα όλα αυτά με πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί η παρουσίαση του κυρίου Ριντόλφη κατέστησε σαφές ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει ολοκληρωμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εγκρίναμε το κονδύλι για την αναπτυξιακή βοήθεια και έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο σχέδιο. Τα, οι τέσσερις πτυχές ε, καλύπτουν πολύ καλά όλους τους τομείς, χρηματοδότηση, αρρωγή και κλίμα επενδυτικό. Πιστεύω λοιπόν πως ε, είναι πολύ καλά δομημένο, όμως πολύ καλά συμπλήρωσε ο κύριος Βαταρά, γιατί μας έδωσε τα κλειδιά των προβλημάτων στην συγκεκριμένη καθημερινή ε, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Πώς θα λυθούν τα τοπικά προβλήματα, τα προβλήματα των κυβερνήσεων που δεν απαντούν, που δεν, δεν λάβουν, στέλνουν τις πληροφορίες εγκαίρως, ε, το ότι οι επενδυτές δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, οι ε, τράπεζες δεν, δεν γνωρίζουν ότι δεν διαβιβάζουν αυτή τη ε, δυνατότητα βοήθειας, ε, την ύπαρξη δυνατοτήτων. Και όταν εμείς γκρίνουμε το, το δεν καταλάβαιναν, δεν ήξεραν ότι υπήρχε εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όντως όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Τώρα, δεδομένως, ε, παρά μάλλον ότι αυτό το μπορεί να καθυστερήσει κάπως τη θέση σε εφαρμογή αυτή η καθυστέρηση, η περιπλοκότητα των χωρών της Αφρικής, αυτό που, που Ωστόσο, είναι σημαντικό είναι ότι τα ωφέλη θα είναι σπουδαία, γιατί θα δοθεί ακόμα μια όθηση σε όλη την αναπτυξή, στην αναπτυξιακή βοήθεια που στέλνουν όλες αυτές οι χώρες που αν χρησιμοποιηθούν μέσα από τις δομές αναπτύσσονται και αυτές, αναπτύσσονται οι τράπεζες, ε, η οικονομία των χωρών, οι κυβερνήσεις. Πιθανότατα είναι πιο εύκολο να δώσουμε την ε, βοήθεια άμεσα στους επενδυτές ε, ή στους διαχειριστές των προγραμμάτων. Όμως είδαμε πως δεν ήταν ε, πολύ αποτελεσματικό και ότι έχει συμβάλει Αντίθετα, σε μεγάλο βαθμό αυτή η επίσημη βοήθεια στην... και αυτό που πρέπει είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πλάνο όπου αναμειγνύονται περισσότεροι φορείς για να το φέρουν εις πέρας, νομίζω πως θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και εφόσον μιλάμε για χρηματοπιστωτικά μέσα, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι δεν σημαίνει πως όλη η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να είναι μέσα στην, στην βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί υπάρχουν project που μπορεί να χρηματοδοτηθούν μόνο με επιδοτήσεις, ενώ υπάρχουν άλλα project που μπορεί να συνδυαθεί η επένδυση με δάνεια να συμπληρωθεί στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Ο πάντως, σε αυτό το στάδιο έχω κάποιες ε, ερωτήσεις και ο κύριος Φερνάντες ρώτησε πότε θα ξεκινήσει. Ε, νομίζω πως είναι καλός τρόπος να, να, ξεκινήσουμε αν και είναι κάπως πιο περίπλοκα στην αρχή τα πράγματα αλλά πιστεύω πως πιο μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει περισσότερο αντίκτυπο το να τα κάνουμε τα πράγματα καλά δεν είναι πάντα εύκολο αλλά πιστεύω πως το κοινό όφελος, το κοινό καλό των Ευρωπαίων και των Αφρικανών και των γειτόνων μας της ε, Ανατολής ε, θα είναι μεγαλύτερο. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Οι συνάδελφοι, αν και είναι προχωρημένη η ώρα, έχουν τίποτα να μας πούνε. Κύριε Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να μάθω για πότε το έχουμε να προχωρήσουμε. να το βάλουμε μπρο. Ο Μάχς, όπως λέμε, το τελευταίο καιρό. Αν ενδιαφέρεται κανείς βέβαια. Και επίσης, Οι υποψηφιότητες για τεχνική βοήθεια προχωράει γιατί έχει και ένα advisory hub το έτσι προχωράει και πώς επίσης το έτσι υπάρχει δυνατότητα για εγγυήσεις σε γείτονες ε, για έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το έχουμε λάβει υπόψη Μήπως μαζί με το έτσι και το Ταμείο Αναπτυξιακής ε, ε, Αϊφόρου Ανάπτυξης μπορεί να φέρει αποτέλεσματα. κύριο Τσέλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στα περισσότερα αφρικανικά κράτη, κατά 90% η οικονομική δραστηριότητα είναι στον άτυπο χώρο της οικονομίας, δηλαδή επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις και θέλω να ρωτήσω πώς θα φροντίσετε έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η οικονομική δραστηριότητα στις, ε, με μικροπιστώσεις πάνω απ' όλα για τις οικογένειες τα λοιπά και πώς θα φροντίσετε έτσι ώστε τα μεγάλα ποσά των πιστώσεων να μην καταλήξουν και πάλι στις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, καταστρέφουν τις δυνατότητες που θα είχε ο τοπικός πληθυσμός με επενδύσεις καταστροφικές στη γεωργία και σε άλλους τομείς. Πώς θα, γίνει, πώς θα ληφθεί επίση με ρήμνα ώστε οι πολίτες των Αφρικανικών κρατών να μένουν στις πατρίδες τους για να δουλέψουν. Και επίσης οι εμπορικές συναλλαγές πώς μπορούν να βελτιωθούν και τελευταίο αλλά πάρα πολύ σημαντικό για τις επενδύσεις ε, και την ενίσχυση της ε, παραγωγής πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Πώς θα, τις, πώς θα την εξασφαλίσετε αυτήν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος και η Ευρώπη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προλαμβάνουν δράση στην Αφρική. Τι γίνεται λοιπόν με όλους τους άλλους ε, παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην Αφρική. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τον Πρόεδρο Γουατάρα. Όντως, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι περιορισμοί μας και κυρίως ε, στον τομέα των χρηματοοικονομικών στις περιοχές αυτές. Έχει δώσει για χρόνια η ΕΤΕΠ ε, επενδύσεις σε διάφορους τοπικούς παράγοντες οι οποίοι δεν έκαναν τις απαραίτητες επενδύσεις και γι' αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα δράσεις με ανοιχτό ε, ανοιχτής αγοράς θα έλεγα ε, γιατί είναι και η ΕΤΕΠ αλλά και πολλοί άλλοι που μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις τους και για να απαντήσω στον κύριο Τσέραρ ταυτόχρονα η πρωτοβουλία αυτή για τις μικρο πιστώσεις είναι ένας από τους άξονες αυτής της δράσης. Διάλογος. Ο διαρθρωμένος διάλογος αναφέρεται και στη δυνατότητα για όλες αυτές τις απαραίτητες δράσεις. Ευχαριστώ την συγκήτρια. είχε κέριο ρόλο στην προετοιμασία του κανονισμού. Βεβαίω περιπλέκονται τα πράγματα με τη συζήτηση, ταυτόχρονα όμω με το One Stop Shop. Όλα τα εργαλεία αυτά λίγο-λίγο εξαφανίζονται, η τεχνική υποστήριξη μπαίνει σε θεματικές ομάδες σε μεγάλα θεματολόγια που έχουν στόχο ακριβώς να εξυπηρετήσουν την ανάπτυξη. Υπάρχουν έργα ανάπτυξης που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από δωρεές βεβαίως. Αυτό δεν αμφισβητείται που δεν είναι. Υπάρχουν ε, οι δυνατότητες για πρόοδο, υπάρχουν τα ζητήματα των πιο ευάλωτων περιοχών, η κρίση, όλα αυτά δεν αμφισβητούνται. Αλλά αυτό που κοιτάμε είναι να, να, να χρησιμοποιούμε στο δυνατόν περισσότερο τα κονδύλια της αναπτυξιακής βοήθειας για να διαφυλάσσουμε ταυτόχρονα και τα κονδύλια των έκτακτων ενισχύσεων, η ανθρωπιστική κρίση κτλ. Χρονοδιάγραμμα είναι το εξή. Ανακοινώνουμε τα πέντε παράθυρα επενδύσεων στην Σύνοδο της Απιτζάν στις 29 στις δε αρχάς ε, του Δεκεμβρίου ανακοινώνουμε την πρόκληση, πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για ε, τελικά χρηματοοικονομικά προϊόντα που θα διατεθούν ως εγγύη στον ιδιωτικό τομέα και αυτό θα μας πάει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου αρχάς Φεβρουαρίου με δύο μήνες ανάλυσης, οικονομικής ανάλυσης από τους ε, τεχνικούς τους επιρρογνώμονες της ε, ΕΤΕΠ αλλά και κοινωνικής οικονομικής ανάλυσης από τις υπηρεσίες επιτροπής από τις αντιπροσωπείες μας στις χώρες και απόφαση, πρώτη συνέπεια θα έλεγα, υπογραφή των χρηματοπιστωτικών μέτρων με την ΕΤΕΠ, την ΆΕΣΥ, την αντίστοιχη γαλλική επιχείρηση και έχουμε και πολλούς άλλους μας έχουν, κάνει, μας έχουν υποβάλει σχέδια μικροχρηματοδότησης που θα μας πάει κάπου στις αρχές Μαΐου, αυτός είναι ο υπολογισμός μας, για να έχουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα των εγγύσεων για τον ιδιωτικό επενδυτή, όπου ήδη κάποιοι επενδυτές έχουν βρει το δρόμο τους προς τα θεσμικά όργανα. Με το One Stop Shop θα τους προωθούμε ταχύτητα και ε, πάντως κάπου τον Ιούνιο περιμένουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα με τα προγράμματα εξωτερική δράσης. Έχουμε περί τι 15 ε, προτάσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προτάσεις για τα πόλεις, για την ενέργεια. Να μας τα πείτε αυτά ότι σας ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν και ζητήματα τεχνικής βοήθειας ε, που σχετίζονται με τον ε, ενεργειακό τομέα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά λοιπόν κατόπιν αιτήματος. Τεχνική βοήθεια, πώς λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό τεχνικής βοήθειας, τρία δις, ένα μεγάλο ποσό τεχνικής βοήθειας, 3 δις λοιπόν σε εκτέλεση ήδη στις χώρες, στις περιφέρειες, τα διάφορα θέματα του θεματολογίου. Όλα αυτά επανοργανώνονται σε μεγάλες ομάδες. Ταυτόχρονα όμως Στηριζόμαστε τεχνική βοήθεια που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας για να ενισχύσουμε τις προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Έτσι γίνεται η οργάνωση και στους ιδιαίτερους τομείς, φερειπίν γεωργία στους επιμέρους τομείς. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη βοήθεια ε, θεσμικών φορέων όπως η ΦΑΟ της Ρώμης, η ΦΑ, το Ταμείο του Γεωργικού, ε, για να βρούμε λύσεις και με τη βοήθεια των παραγόντων, των φορέων επιτόπου. Για τον κύριο Τσέλερ μερικές φορές είναι άτυπη αυτή η οικονομική δραστηριότητα. Βέβαια δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτήν την κατάσταση ως μια μόνιμη κατάσταση. Πρέπει δηλαδή να κοιτάμε να βοηθήσουμε να ε, οριμάσει αυτή η οικονομική δραστηριότητα. Υποστηρίζουμε τις μικρο ε, οικονομίες και τις πολύ πολύ μικρές βέβαια ε, τοπικές επιχειρήσεις αλλά πρέπει να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν και μεγαλύτερες επιχειρήσεις με μια θετική δυναμική. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να μείνουν στις χώρες οι επενδύσεις. το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε με τους κανόνες για τις επενδύσεις. Εάν υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τηρούνται βεβαίως από, τα θεσμικά, από τους θεσμικούς φορείς και πρέπει να φροντίσουμε τα ωφέλη να στοχεύουν στη δημιουργία θέσεων εργασία στο τοπικό επίπεδο. Πώς θα βελτιώσουμε τις εμπορικές σχέσεις. Έχουμε συζητήσει επί μακρόν, πιστεύω, τις συμφωνίες οικονομικής ε, εταιρικής σχέση. Πρωτόκολλο της Επιτροπής του ΛΟΜΕ και το καθεξής. Έχει γίνει συζήτηση για πολλά χρόνια. Δεν έχουμε φτάσει να την ολοκληρώσουμε, αλλά αν το καταφέρουμε θα τους ενισχύουμε ιδιαίτερα το δυναμικό τους και βέβαια το, η δημογραφική πρόκληση για την οποία έγινε λόγος νωρίτερα σημαίνει μια μεγάλη ευκαιρία για την αγορά. Δεν είναι μόνο εκμετάλλευση από πλευρά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αλλά και δυνατότητες για τις τοπικές και περιφερειακές αγορές. Η Αφρική, ξέρετε, εισάγει και πολλές τροφές, πολλά τρόφιμα, δεν γίνεται κατεργασία, δεν ε, προσφέρεται τη θεμενή αξία. Και αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, τον ε, Διευθυντή Πλανήτης και Ευημερία. 12 και 40 τα καταφέραμε. Μπράβο σας και ευχαριστούμε και τους δερμηνείς που αντέξανε. Ακρόαση άκρο συναρπαστική. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους και όσους συνάδελφους άντεξαν και αυτοί ως το τέλος. Μια ακρόαση γεμάτη υποσχέσεις. Δεν φαντάζομαι να στα έκανες άλλο στο λόγο. Χαίρετε. 12, 2 και 30 συνεχίζουμε. Με τον Hans Geier στο ρόλο του Προέδρου. la Skills Week, qui est une façon d'apporter une réponse au chômage des jeunes en Europe. Et j'ai noté que parmi les éléments de développement en Afrique, il y avait aussi l'apprentissage